Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε παρακαλώ με τις ψηφοφορίες. Μία γνωμοδότηση έχουμε μόνο να ψηφίσουμε του Derek Vaughan για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους. Αλλά πρώτα ας ελέγξουμε τα μηχανήματα. Βάλτε παρακαλώ τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας για να ελέγξουμε αν λειτουργούν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 ψηφί. Okay. Well, machine shows that 31 cards were... Βλέπω ότι 32 κάρτες μπήκαν στις συσκευές, αλλά μόνο 30 ψήφισαν. πάντως το σύστημα λειτουργεί, οπότε ας περάσουμε στην ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8, ποιος είναι υπέρ, υπέρ της 8 κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 8. Μήπως βάλετε λάθος κάρτα. It doesn't work. So, so we... No. No, but, uh, but his card is not working, so that's why I'm... It's fine? Yeah. Yes, Victor, you... Somebody voted for you. Okay. Victor, μάλλον κάποιος άλλος ψήφισε. Για σένα, εν πάση περιπτώσει, εγκρίθηκε ομόφωνα η τροπολογία. Οκτώ. Αποκλείεται όμως, αφού ήσασταν κατά, πώς ομόφωνα. Ψηφίζουμε το, την 8. Και η μισή ήσασταν κατά, τώρα ξαφνικά όλοι γίνεται υπέρ. Εν πάση περιπτώσει, 29 υπέρ. εγκρίνεται η τροπολογία 8. Δεν χρειάζεται να επαναληφθεί η ψηφοφορία, είναι σαφέ ότι ψηφίστηκε. Η τροπολογία 9, ποιο είναι υπέρ, κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 16 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 16 Yeah, which, uh, the vote is Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 20 υπέρ, 13 κατά. Τροπολογία 17. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 17. Εγκρίνεται με 18 υπέρ, 15 κατά 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές ασαφές το αποτέλεσμα. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 15 υπέρ, 18 κατά και τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 42, ποιος είναι υπέρ, κατά άποχες απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά άποχες εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 ψηφοφορία κατά τμήματα πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Μάλλον απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα, της 53. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, 19 κατά 14 υπέρ. 54 ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονικό τρόπο άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται ομόφωνα η γνωμοδότηση έτσι λαμπρά συγχαρητήρια στον εισηγητή μας τον κύριο Βόν Ε, Ωραία συνάδελφοι. Θα θυμάστε ότι χθε συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε σήμερα το πρωί την ε, απογευματινή συζήτηση για το νέο πακέτο του κανονιστικού πλαισίου. Θα ήθελα καταρχήν να σας ε, ενημερώσω εν συντομία ε, τι είπαμε στην ομάδα εργασία, παρουσία των συντονιστών και των εισηγητών. Εκεί λοιπόν συμφωνήσαμε με βάση την απόφαση της Επιτροπής της 5 ε, η Οκτωβρίου η ομάδα εργασίας να συντονίσει πλέον, να συντονίσει πλέον ολόκληρη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ομάδα εργασίας για να συνεννοούμαστε με τους συντονιστές, γιατί συμφωνήσαμε ότι θα χρειαστούν πολλές συντονιστικές προσπάθειες για τις διαπραγματεύσεις, γιατί σίγουρα ο Γενικός Κανονισμός σχετίζεται άμεσα με τους επιμέρους κανονισμούς για τα επιμέρους ταμεία, οπότε θα χρειαστεί μεγάλο συντονισμός και αυτό το αντιλήφθηκαν οι εισηγητές και συμφώνησαν να χρησιμοποιηθεί αυτή ε, η ομάδα ως πλατφόρμα συντονισμού. Κάτι άλλο που συμφωνήσαμε είναι να τη χρησιμοποιήσουμε και για διευκρινιστικές ε, συναντήσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Πάντως όλες οι αποφάσεις και όλες οι συζητήσεις που θα γίνουν ε, θα μεταφέρονται και στην Επιτροπή εδώ. Κάθε δύο μήνες αποφασίσουμε να έχουμε συζήτηση για τους επιμέρους κανονισμούς και αποφασίσαμε και για τις προθεσμίες ένα χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα του Συμβουλίου και της Επιτροπής, αποφασίσαμε να διεκπαιρεώσουμε την όλη διαδικασία μέχρι τα τέλη του 2012. Βέβαια, είπαμε ότι υπάρχει άρρηκτος δεσμός μεταξύ του δικού μας ρυθμιστικού πλαισίου για το οποίο είναι συνεισηγητές η Κωνσταντσα Κρέλ και ο Λάμπερτ. Βέβαια, ο Λαμπέρ απουσίαζε, αλλά τον κάλυψε η Κωνσταντζ, γι' αυτό λέω, συμφωνούν οι δύο συνεισηγητές. Είναι λοιπόν ε, δεδομένη η σπουδαιότητα του γενικού κανονισμού για τους επιμέρους κανονισμούς. Τα περισσότερα θέματα ε, αναφέρονται εκεί οριζόντια, οπότε συμφωνήσαμε για στενή συνεργασία και με τις υπόλοιπες επιτροπές που είναι αρμόδιες για τα λοιπά ταμεία, ιδιαίτερα την Επιτροπή Απασχόλησης αλλά και την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη νομική μορφή, ιδιαίτερα για τη συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Μια άλλη πρόταση είναι η επόμενη γενική συζήτηση επί των σχεδίων εκθέσεων να γίνει την Άνοιξη. Κατά πάσα πιθανότητα τον Απρίλιο. Αλλά δεν ορκιζόμαστε κιόλα. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτά εξετάσαμε και αποφασίσαμε χθες στην ομάδα εργασίας. Πάντως ε, η παράκλησή μου είναι όλες ε, οι αποφάσεις και οι τακτικά συζητήσεις να μεταφέρονται και εδώ στην Επιτροπή μας. Επανερχόμαστε τώρα στη χθεσινή συζήτηση του απογεύματος. Θα δώσω το λόγο στους ε, συνεισηγητές του Γενικού Κανονισμού να κάνουν κάποια σχόλια, αν θέλουν. Δεν είναι υποχρεωμένοι όμως. Ο Λαμπέρτ ή η Κωνσταντσα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. χθε είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε νέες πληροφορίες, αλλά τελικά είχαμε τόσε πολλές που δεν ξέραμε ποια ήταν τα βασικά. Χτες, λοιπόν, μοιράσαμε το άτυπο έγγραφο εργασία με τα 11 σημεία που μπορεί τώρα να γίναν 12. Εν πάση περιπτώσει αυτά είναι τα οριζόντια θέματα που θέλουμε να αναφέρουμε. Η αίσθησή μου είναι πως ε, η πρώτη συζήτηση νομίζω σας ε, είχε και σας λάβει υπόψη, δεν είναι τόσο διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει ένα λογικό πλαίσιο λοιπόν νομίζω εδώ, οπότε σε εργαστούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ίσως είναι λογικό να έχουμε στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μία συζήτηση για κάποια από τα βασικά ζητήματα. Ίσως κάποια να είναι τόσο σημαντικά, εάν μιλάτε π.χ. για μακροαιρεσιμότητα, αρχίσουμε να, χτυπιόμαστε και να μην πάει πουθενά η πρόταση. Οπότε θα το αποφασίσουμε αυτό αργότερα, όταν θα φτάσουμε στις πτυχές της πολιτικής ε, της ε, μακροαιρεσιμότητας αλλά υπάρχουν άλλα θέματα ε, όπως η ευελιξία, όπως τα εταιρικά αυτά συμβόλαια που συζητήσαμε χτες. Ίσως λογικό είναι να αφαιρέσουμε τέσσερα σημεία και να σας τα στείλουμε. Όχι να αφαιρέσουμε, αλλά να ασχοληθούμε, με τέσσερα σημεία σε βάθος. Οπότε να πούμε ότι κάνουμε μια συζήτηση και μετά θα φτάσουμε στις τροπολογίες και τα λοιπά. Γιατί σε τελική ανάλυση θα είναι τεράστιο αυτό το θέμα. Για να υπάρχει και συνεργασία. Βεβαίως γιατί υπάρχουν και πολιτικές ομάδες και δεν θα επιτύχουμε ποτέ το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει ο Πρόεδρος μία ακόμα παρατήρηση. Δεν είμαστε μόνοι ως ε, Κοινοβούλιο. Αυτή την εβδομάδα υπάρχει άτυπη υπουργική ε, διάσκεψη στο Πόσναν και ξέρουμε πως ε, και το Συμβούλιο βήμα-βήμα ασχολείται με κάποια κομμάτια αυτού του κανονισμού. Οπότε κάποια, η διαδικασία αυτή ε, εξελίσσεται και κάποια πράγματα αλλάζουν και στο Συμβούλιο. Οπότε η ομάδα αυτή εργασία βεβαίω δεν λαμβάνει καμία ευθύνη τη Επιτροπή μα, αλλά είναι κάτι το σημαντικό. Οπότε να μην ξαναξεκινήσει η όλη συζήτηση. Βεβαίω αναμένω να δούμε τι ε, θα προκύψει, ίσως λάβουμε το λόγο, να πω και το εξής. Εγώ και η Κωνσταντζα θέλουμε να είμαστε εισηγητές. Ε, υπάρχουν δύο εισηγητές επί του θέματος. Δεν είμαστε συνεισηγητές, να μας λέτε εισηγητές. Γιατί μετά λένε που είναι ο συν ο δικός σου. Ε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Κωνσταντζα έδωσε ένα καλό παράδειγμα. Η Κωνσταντζα είπε εγώ είναι δικιά μου η γνωμοδότηση, δικιά τη είναι έτσι. Δεν είναι ότι πηγαίνουμε μαζί και στην τουαλέτα, αλλά θα τα καταφέρουμε. Ε, Καλώς. Ε, ποιος ε, είπε συνεισηγητή. Ποιος σε αποκάλεσε συνεισηγητή. Εγώ τουλάχιστον ποτέ. Αλλή μόνο. Ωραία, ελπίζω να, συμφωνήσουμε λοιπόν ότι στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Βέβαια είναι κοντά στα Χριστούγεννα, αλλά ελπίζω παρόλα αυτά να έχουμε σημαντική προσέλευση. Έχουμε το θέμα της συγκέντρωσης των συμβάσεων εταιρική σχέσης ε, και άλλα επιμέρους ζητήματα, αλλά πιστεύω ότι αν οι εισηγητές των επιμέρους ταμείων ασχοληθούν με το θέμα αυτό θα το καταφέρουμε. Πάντως αυτό που υπήρχε αρχικά στο γενικό κανονισμό έχει περιληφθεί και στους επιμέρους κανονισμούς για τα ταμεία. Ορισμένα θέματα λοιπόν που επηρεάζουν και εσάς και το περιεχόμενο της δικής έκθεσης περιλαμβάνονται και στο γενικό κανονισμό. Οπότε πρέπει να είστε έτοιμοι για τη συζήτηση υπό το πρίσμα φυσικά του κανονισμού που επεξεργάζεστε εσείς. Α είμαστε συγκεκριμένοι. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για τον γενικό κανονισμό, θα έχουμε δύο-τρία συγκεκριμένα θέματα. Να είστε προετοιμασμένοι. Ωραία, περάμε τώρα σε άλλε εκθέσει. Καταρχήν θα ήθελα να προτείνω το εξή. Έχουμε μία ώρα και 20 λεπτά περίπου για όλου του κανονισμού. Θα προδώσω πρώτα το λόγο στους συγητές να παρουσιάσουν τις εκθέσεις τους και μετά θα ακούσουμε τους κοιόδης συγητές και τους υπόλοιπου ε, ομιλητέ. για να μην αφήσουμε ε, εκτός συζήτησης καμία έκθεση και κανένα κανονισμό. Χρόνου φίδου, αλλά φυσικά θέλουμε μεστή παρουσίαση. Ε, η πραγματική πρόκληση είναι ότι υπάρχουν τα ίδια στοιχεία σε όλους τους κανονισμούς. Και χωρίς να εξειδικεύσουμε τα στοιχεία γενικά, θα έχουμε προβλήματα και με τους άλλους κανονισμούς. Για παράδειγμα, να τονίσω κάποια από τα στοιχεία που έχουμε εδώ. Πρέπει να φύγω. Ε, χθες δεν είχα την ευκαιρία να λάβω μέρος ε, στη συζήτηση, αλλά είναι σημαντικό για σήμερα. Πρώτον, πρώτη, πρώτο ζήτημα. Η Επιτροπή ως συγγραφέας του κειμένου, τι θα γίνει με τους θεματικούς στόχους. Αυτό έχει οριστικοποιηθεί ε, είναι ένα κείμενο του κανονισμού που θα τροποποιηθεί. Γιατί αν έχει οριστικοποιηθεί, είναι μια σαφής μετάφραση του, 20, ε, του 2020. Ή πρέπει να το επεξεργαστούμε περισσότερο. Ε, μετά έχουμε το επόμενο, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχουμε το εξή. Έχουμε τις συνέπειες για τις προτεραιότητες των επενδύσεων. Αυτές όμως μεταφράζουν τους θεματικούς στόχους. Χωρίς τους θεμα... Αφού οριστικοποιηθούν πρώτα οι στόχοι, θα χρειαστεί να τροποποιηθούν και οι προτεραιότητες της επενδύσης. το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι αρκετά μικρό, αλλά επειδή συνδέεται με τους άλλους κανονισμούς, περιπλέκεται το ζήτημα. Έχουμε τον κατάλογο των δράσεων, των επιλέξιμων και των μη επιλέξιμων. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν θέλω να πω στις λεπτομέρειες γιατί έχουμε τη δυνατότητα στήριξης από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, θετικό, πρέπει να το στηρίξουμε. Αλλά υπάρχουν και πράγματα που δεν πρέπει να στηρίξουμε. Ε, αυτά που δεν πρέπει να στηρίξουμε είναι πολύ συγκεκριμένα. Δεν είναι γενική κατηγορία πράξεων, για παράδειγμα πυρηνική ενέργεια, αλλά υπάρχει και η παραγωγή του καπνού. Θέλω να ρωτήσω, γιατί ο καπνός, γιατί υπάρχει ο καπνός στον κατάλογο, γιατί όχι η τα πρόβατα ή οι μπανάνες. Εντάξει, ξέρω γιατί είναι σημαντικός ο καπνός, αλλά είναι ο μόνος τύπος παραγωγής που πρέπει να απαγορευτεί. Υπάρχουν πολλές περιοχές στην Ευρώπη όπου υπάρχει πολύ σημαντική παραγωγή καπνού και καλλιέργεια καπνού. <clears throat> τι είναι επιλέξιμο λοιπόν και τι δεν είναι επιλέξιμο. Το ερώτημα σε σχέση με τη θεματική ε, συγκέντρωση. Όπως ξέρετε, ε, υπάρχουν και ε, πράγματα που λαμβάνονται από το γενικό κατάλογο, τρία συγκεκριμένα. Και φυσικά ο γενικός κατάλογος είναι πολύ σημαντικό και είναι και πολύ διάσημο αυτό το 80%. 80% για τις πιο ανεπτυγμένε περιοχές. Και αν θυμάστε την πρόταση των δύο εισηγητών, όχι συνεισηγητών, αυτοί ε, είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα έβαζαν κατά μέρου συγκεκριμένου πόρου και τώρα μιλάμε ήδη για 80% για του τρει θεματικού στόχου, του οποίου παίρνουμε από του γενικού στόχου. Νομίζω πρέπει να διευκρινιστούν αυτά. Πρώτα, να οριστικοποιηθούν οι θεματικοί στόχοι. Δεύτερον, αυτά τα τρία, αυτοί οι τρει τομεί, τα τρία θέματα και, εν πάση περιπτώσει, θα ε, ε, αφιερώσουμε συγκεκριμένου πόρου για συγκεκριμένου τομεί ή όχι. Υπάρχει και μια έντονη αστική συνιστόσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το, η οποία συνιστόσα είναι μεν πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά είναι εξίσου ασαφής. Ασαφής λέω. Με την ευκαιρία θα ήθελα να τονίσω και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό γιατί τα κράτη-μέλη θα αρχίσουν να ε, ε, ετοιμάζουν τις συμβάσεις τώρα. Χθες όμως στις Βρυξέλλες άκουσα ότι η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ των κρατών μελών και των Βρυξελών, που δεν είναι αλήθεια. Λάμπερτ και Κωνσταντς, ε, εσείς λέτε στα κείμενά σας ότι η σύμβαση θα ε, υπογραφεί μεταξύ, μεταξύ των κρατών μελών και της ε, Επιτροπής. Ούτε αυτό είναι αλήθεια. Μεταξύ κυβερνήσεων υπογράφονται αυτές οι συμφωνίες. Πρέπει να δούμε λοιπόν το σύστημα υλοποίησης. Θα πρέπει να έχουμε έναν κατάλογο με τις πόλεις οι οποίε θα έχουν αυτή την ολοκληρωμένη αστική δράση. Ε, η Επιτροπή λέει περίπου 20. Ε, το φαντάζομαι για τη Γερμανία, εντάξει, αλλά το Λουξεμβούργο τι γίνεται. 20 πόλεις στο Λουξεμβούργο. Ε, κατάλογος πόλεων, λοιπόν. Κατά συνέπεια, και σας προτείνω να διαβάσετε το κείμενο, γιατί αν το πάρουμε στην κυριολεκτική του έννοια, σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη επιλέγουν κάποιες λειτουργικές περιοχές ονομάζεται αυτό ολοκληρωμένο ολοκληρωμένη αστική δράση. Πρέπει μετά να καταρτιστεί ολοκληρωμένη στρατηγική. Αν καταρτιστεί ολοκληρωμένη στρατηγική, ε, μπορούν να προγραμματιστούν ολοκληρωμένες αστικές δράσεις. Υπάρχει και ένα περίφημο καινούριο στοιχείο. Πώς ονομάζεται, ε, πώς το λέμε, πώς το λέμε, πώς πρωτοβουλία εδαφική για το 5%. Το 5% λοιπόν από ό,τι φαίνεται, και αυτό έχει να κάνει για τις ε, ολοκληρωμένες αστικές δράσεις για τον κατάλογο των πόλεων, σημαίνει μόνο για τις πόλεις που είναι στον κατάλογο το 5%. Και στη συνέχεια οι, οι πόλεις αυτές θα πάρουν μέρος και στην αστική πλατφόρμα. Όλες οι πόλεις της Ευρώπης μας ρωτάνε ποια πόλη θα είναι στον κατάλογο, ποιες πόλεις θα είναι στον κατάλογο, τι είδους πόλεις κτλ. λοιπά Και αυτό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Λοιπόν, πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι εννοεί με αυτές τις προτάσεις. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια λογική αλληλουχία Πολύ συχνά οι πόλεις στην Ευρώπη αναρωτιούνται, είναι 5% για τις αστικές ε, δράσεις, τι είναι 5% είναι τίποτα δεν είναι. Ε, αν το 5% αφορά τα ολοκληρωμένα αστικά προγράμματα, αυτό σημαίνει ότι είναι ένα είδος πιλωτική εφαρμογή κτλ. κτλ. Ε, πρέπει να το κάνουμε λοιπόν. Ε, πρέπει να αναρωτηθούμε τι είναι από πίσω, ποια είναι η, η ιδέα, η κινητήρια. Αν εδώ θέλουμε μια πιλωτική εφαρμογή για μια, έναν κατάλογο πόλεων για να καταρτιστούν αυτά τα ολοκληρωμένα σχέδια και αφιερώσουμε και ένα 5% με μια ειδική μεθοδολογία, αυτό είναι λογικό. Εντάξει, τι εννοεί η Επιτροπή. Στη συνέχεια, ο κατάλογος με τους δείκτες, πολύ σημαντικός, γιατί αυτό είναι συνέπεια των θεματικών στόχων, των προτεραιοτήτων στις επενδύσεις και των... μετά έρχονται οι δείκτες. Και το θέμα είναι, οι δείκτες είναι στο παράρτημα. Μπορούμε να τροποποιήσουμε και τον κατάλογο των δικτών. Μπορούμε να προτείνουμε καινούριου δείκτες. Μπορούμε να μεταβάλουμε τους υπάρχοντες δείκτες όπως και το κείμενο του κανονισμού. Ε, αυτό όλο ε, απαιτεί πληροφορίες. Είναι πολύ σημαντικό. Πρόκειται για ένα νομικό κείμενο. Λοιπόν, θεματική στόχη. Είναι το νομικό κείμενο ή είναι η Πληροφορίε για το παράρτημα του νομικού κειμένου. Τι συμβαίνει με τι συμφωνίε για τι εταιρικέ σχέσει, Ποιοι είναι οι εταίροι. Αυτό είναι ζωτική σημασία. Και όσο αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή ανάπτυξη, τι θα γίνει με τις επιλέξιμε δαπάνε. Ποιε είναι. Θα έχουμε πολλέ συνομιλίε με την Επιτροπή στο μέλλον. Γιατί λοιπόν αναφέρεται ο καπνό, Τι το τόσο ιδιαίτερο έχει η καλλιέργεια του καπνού. Ε, ολοκληρώνω. Είμαι λογικός. Και βέβαια, η, η αφιέρωση συγκεκριμένων πόρων, η αστική συνιστόσα και φυσικά οι δείκτες. Αυτά θα πω προς το παρόν. Είναι πολύ σημαντικό το ETPA, το ΕΤΠΑ, αλλά δεν μπορούμε να ε, συζητούμε για τις λεπτομέρειες χωρίς να ξέρουμε το γενικό πλαίσιο. Έχουμε την εδαφική συνεργασία ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αν δεν λύσουμε τα προβλήματα αυτά θα παγιδευθούμε. Προς το παρόν είμαι αισιόδοξο γιατί το ΕΤΠΑ είναι πιο ευέλικτο. Ταυτόχρονα όμως για την αφιέρωση συγκεκριμένων πόρων 80%, 50%, ε, εκεί θα γίνει ο μεγάλος καυγάς. 80%, 60% είτε θα κάνουμε την πολιτική πιο ευέλικτη ή θα διοχετεύσουμε ήδη από τώρα τους πόρους. Ε, υποθέτω ότι αυτό θα είναι το πιο δύσκολο ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα καλωσορίζω τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, τον Νίκολας Μάρτιν. Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Μποστινάρου, να πω το εξής. Νικόλα, θα θέλαμε να σε ακούσουμε ε, μετά τους συναδέλφους να απαντήσει διάφορες ερωτήσεις, αλλά να πω στο Γιάννη. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα εκτός από τις επεξηγηματικές δηλώσεις. Οπότε είμαστε υπεύθυνοι για το τι θα προτείνουμε, αλλά ο ρόλος μας δεν είναι μόνο να ζητάμε διευκρινήσεις, αλλά να αλλάζουμε και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Σας ενθαρρύνω για μην νομίζετε ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε τίποτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, απλά ε, για να μην νομίζετε ότι είναι προκλητικές οι ερωτήσεις μου. Όχι, όχι, σας ξέρω εδώ και καιρό, ξέρω ότι είστε προκλητικός. Βίκτορ Μποστινάρο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ούτε εγώ θέλω να είμαι ούτε προκλητικός ούτε προβοκάτορας. Δύο σχόλια σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Όλμπεριχτ. Υπάρχει η άποψη πως με κάποιο τρόπο η πολιτική συνοχή είναι τώρα ο βασικός μοχλός στρατηγικής του 2020 σε όλα τα έγγραφα από την Κομισιόν φαίνεται πως η πολιτική συνοχής έχει φύγει από το βασικό της στόχο ε, που είχε όταν ε, ξεκίνησε. Κατόπιν για τη μακροοικονομική σταθερότητα είναι προφανές πως ε, η ομάδα μας, αλλά όχι και άλλες, και όχι μόνο η ομάδα μας, και άλλες πολιτικές ομάδες ξέφρασαν ανησυχίες για το να μπουν μακροοικονομικές αίρεσιμότητες στην πολιτική συνοχή. Τρίτον, όταν υπάρχει αυτό το αποθεματικό το 5% συν ε, ένα ανώτατο όριο, συν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ε, του μέσου του ευρώ, θα δείτε πως στην πράξη η πολιτική συνοχής χάνει ένα πολύ σημαντικό ε, ποσό που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Τέλος, πράξη κατεξιοδότηση. Μας το είπαν χθες. Όπως ξέρετε κύριε Γενική, κύριε Γενική Διευθυντά, γιατί Μάρτιν και στο Συμβούλιο ήταν κατά των πάρα πολλών πράξεων κατεξιοδότηση. Και ξέρετε πως αυτό δημιουργεί προβλήματα στο Συμβούλιο και απογοήτευση και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Τώρα, για το Μέσο συνοχή, θα αναφερθώ σε τρεις σημεία. Πρώτον, μιλάμε για το μέσο σύνδεσης της Ευρώπης, ε, γιατί το οποίο πλέον είναι 68 δισεκατομμύρια, σχεδόν το ίδιο με το Ταμείο Συνοχής. Αλλά, γιατί μας στέλνει εδώ πέρα ένα έγγραφο η Κομισιόν, το οποίο είναι, σας το λέω ξεκάθαρα, ασαφές τίποτα το συγκεκριμένο. Κάποιες βασικές ερωτήσεις λοιπόν για τη φιλοσοφία, για την κοινή διαχείριση και η κεντρική διαχείριση του μέσου ε, σύνδεσης της Ευρώπης. Πράγματα τα οποία κάπως συγκρούνται. Δεύτερον, είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι τα κριτήρια για να φύγουν τα 10 δισεκατομμύρια από τα κράτη-μέλη να πάνε στην κεντρική διαχείριση και μετά να αποφασίσουμε ποια είναι τα καλύτερα έργα. Γιατί είναι σαφές πως ε, θα είναι πάνω από ένα κράτος μέλος, θα είναι δύο ή και περισσότερα. Με ποια κριτήρια πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό, αλλιώ. θα έχουμε μάχη και στο Κοινοβούλιο και άλλη μία μάχη στο Συμβούλιο. Και τέλος τι γίνεται με τους εργολάβους όταν μιλάμε για μεγάλα νούμερα, πολλά λεφτά, είναι προφανές πως θα έχουμε προβλήματα και καλό είναι να αποφύγουμε περαιτέρω απογοητεύσεις και να μην υπονομεύουμε τη δυνατότητα συμφωνίας. Και ελπίζω πως ε, μετά την παρουσίαση της Κομισιόν θα μπορούσαμε ίσως να ξεκαθαρίσουμε λίγο την κατάσταση. Δεύτερον, for, ε, για τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το Ταμείο Συνοχής ε, για να πληρώσουμε για τη ρήπανση όταν δεν πληρώνει ο ρηπαίνων λόγω της πολύ μεγάλης ρήπανσης. Εάν επί της αρχής είμαι υπέρ, στην πράξη θέλω να σας πω, κύριε Μάρτιν, πως δεν έχουμε ξεκάθαρη απάντηση για τα κριτήρια που υπάρχουν σήμερα, δηλαδή στρα, ε, αξιολόγηση ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πράγματα τα οποία δεν είναι ουδέτερα, είναι ξεκάθαρο πως δεν μπορούμε να δώσουμε πράσινο φως για αυτή τη δυνατότητα, γιατί θυμηθείτε στην Ουγγαρία για τη ρήπανση προκάλεσε μια ιδιωτική εταιρεία ή η κυβέρνηση έβαλε πρόσφατα 500 εκατομμυρίων ευρώ, τεράστια, για να αποτραπεί ακριβώς η ρήπανση και για να μην υπάρχει δυνατότητα να μην πληρώσει. pollution and then he will also be able to pay the pollution αποτρεπτικό ρόλο δηλαδή παίζει, αλλά και να πληρώσει βεβαίω για τη ρήπανση. Δεν ξέρω γιατί να χρησιμοποιηθεί αυτό το ταμείο για αυτό το λόγο, όταν υπάρχει περιβαλλοντική πολιτική και θα πρέπει βεβαίω να έχει προληπτικό ρόλο. Και η τελευταία μου πρόταση αφορά την δυνατότητα πρόσβαση στο Ταμείο συνοχή για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα στον τομέα των... της στέγασης τον ε, υφιστάμενο κανονισμό είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά έχοντας υπόψη ε, την κλιματική αλλαγή, μετά εκτιμώντας το ότι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα θα κάνει την ενέργεια προσβάσιμη στον κόσμο που πληρώνει την κρίση, μπορεί να θεωρήσουμε αυτή τη δυνατότητα όχι μόνο φιλική προς το περιβάλλον, δηλαδή εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά επίσης μείωση του αερίου και θα αυξήσει επίσης το ποσοστό της ανανεώσιμης ενέργειας ε, στο σύνολο της παραγωγής και της κατανάλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους στόχους στρατηγικής του 2020. Αυτές είναι οι βασικές μου ανησυχίες και είμαι πεπισμένος πως ε, δεν είναι μόνο δικές μου, αλλά και περισσότεροι συνάδελφοι έχουν την ίδια άποψη και είμαι πεπισμένος πως με τη στενή συνεργασία μεταξύ πολιτικών ομάδων και ημών Κομισιών και Συμβουλίου θα αποφύγουμε αιματηρές μάχες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Βίκτορ. Η ε, Ρίκα Μάνερ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ασχολούμαι με το στόχο της εδαφικής συνεργασίας στο ΕΤΠΑ. Πρώτη φορά που περιλαμβάνεται αυτός ο στόχος στον κανονισμό. Έχω κάποια γενικά σχόλια για τον κανονισμό που μου κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από ένα περίπου μήνα. Όπως θα ξέρετε και όπως προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στην εσωτερική αγορά, αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις που μερικές φορές είναι δύσκολες. Ε, γιατί μερικές φορές ε, οι προκλήσεις ξεπέρνουν τα περιφερειακά και εθνικά σύνορα, γι' αυτό και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ε, που είναι, έχει πια πανευρωπαϊκή διάσταση είναι πολύ σημαντικός και αυτή είναι η βάση και του σχετικού κανονισμού. Πώς μπορούμε λοιπόν να υλοποιήσουμε τους στόχους αυτούς ε, από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για να αντιμετωπίσουμε τα κοινά προβλήματα όπως είναι περιβαλλοντικά, διασυνοριακή χρήση νοσοκομείων, ανταλλαγή εμπειριών, άνοιγμα της βιομηχανίας και του εμπορίου με διαφανή τρόπο κτλ. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις και τα σχόλια ε, περιλαμβάνονται και στο σχετικό κανονισμό. Πολύ σημαντικά λοιπόν όλα αυτά και... Ah, okay. It's based also... ε, ο νέος κανονισμός σε μεγάλο βαθμό ε, μοιάζει με το προηγούμενο ΕΤΠΑ, του προηγούμενου πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Χρειαζόμαστε λοιπόν εδαφική συνεργασία πανευρωπαϊκή και αυτή η εδαφική συνεργασία ε, χωρίζεται σε τρία προγράμματα στο νέο κανονισμό ε, που καλύπτουν τη διασυνοριακή, την εθνική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία. Το πρώτο θέμα ήταν η διασυνοριακή συνεργασία. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τέτοια είδο διασυνοριακά σχέδια των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Έχουμε τέτοια στη Γερμανία και Πολωνία για να επιληθούν προβλήματα υποδομών μεταξύ των δύο χωρών. Σχεδόν όλα τα σύνορα καλύπτονται από τέτοιου είδους προγράμματα εδαφικής συνεργασίας. Αυτή η διασυνοριακή συνεργασία αποτελεί ε, οριζόντιο στόχο. Γι' αυτό και προβλέπεται και σχετικός προϋπολογισμός. Και το περιλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο νέο δημοσιονομικό, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά την ε, δαφική συνεργασία στο νέο κανονισμό, ε, έχει διακρατικό χαρακτήρα και προσπαθεί να, να προωθήσει την ε, συνεργασία μεταξύ περιφερειών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις, στην περιοχή της Βαλτικής, στις Άλπεις. Επίσης έχουμε συγκεκριμένες περιοχές εδαφικής συνεργασίας. Και τέλος το μικρότερο τμήμα του κανονισμού αφορά την τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας που στόχο έχουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για καινοτομία, ενεργειακή αποδοτικότητα, ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Η ιδιαιτερότητα αυτών των προγραμμάτων έγκυται στο ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν ακόμη και εκτός Ένωσης. Και η Νορβηγία και η Ελβετία συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Τώρα, για το συγκεκριμένο κανονισμό, τι θα αλλάξει ο κανονισμό σε περίπτωση φυσικά που ε, εγκριθεί η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιληφθεί στο κοινοτικό κεκτημένο. Καταρχήν, ε, θα, θα πρέπει οι εταίροι αυτών των προγραμμάτων να συμφωνήσουν συγκεκριμένα τι προγράμματα θα χρηματοδοτήσουν και να θεσπίσουν συγκεκριμένους στόχους. Κάτι αντίστοιχο ακούσαμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ίδιο σύστημα ακολουθεί και ο κανονισμός για την εδαφική συνεργασία. ETC. Τα σχέδια αυτά και τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται φυσικά με τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών πολιτικών και των στρατηγικών ε, προκειμένου φυσικά να ληφθεί υπόψη και ο στόχος ενεργειακής αποδοτικότητας και να βρεθούν και κάποιες συνέργειες μεταξύ των περιφερειών. Ε, όλα φυσικά αυτά εντάσσονται στους στόχους της στρατηγικής του 2020 και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας υπάγονται εκεί. Η σχετική νομοθεσία θα τονώσει ιδιαίτερα την ε, συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών και θα προσπαθήσει να ελαφρύνει το γραφειοκρατικό και διοικητικό άχθο για του διαχειριστέ των προγραμμάτων. Αυτό είναι ένα νέο τμήμα του κανονισμού, γιατί γνωρίζουμε ότι και στα προγράμματα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, ETC, προβλέπεται έντονη γραφειοκρατία. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένε προτάσεις για την απλοποίηση των διατυπώσεων. Τέλος, προβλέπεται περισσότερη ελαστικότητα για τα διάφορα κονδύλια του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και οι επενδύσεις αυτές φυσικά θα πρέπει να ευνοούν ιδιαίτερα τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Είναι σαφές τώρα το ζήτημα του ελέγχου και της λογοδοσίας για τη χρήση των κονδυλίων μεταξύ των εταίρων. Ένα σημείο του κανονισμού που με βρίσκει ιδιαίτερα σύμφωνη είναι αυτή, αυτό το καταποκοπή ποσό για το 50% για τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Χρησιμοποιείται αυτό το 50% αυτό το καταποκοπή ποσό για τεχνική αρρωγή κυρίω. Και αυτός είναι και ένας τρόπος για να μειωθεί η γραφειοκρατία. Οι πρώτες αντιδράσεις ε, για το νέο κανονισμό ήταν σχετικά θετικές, υπήρξε μάλλον ικανοποίηση και φυσικά τηρούμε τους κανόνες της προηγούμενης περίοδου του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Πάντως πιστεύουμε ότι με το νέο κανονισμό θα έχουμε κάποια πλούστευση των διαδικασιών. Κάποια άλλα σαφή σημεία στον κανονισμό θα ήθελα να επισημάνω τώρα. Καταρχήν, το θέμα το, της θεματολογίας των προγραμμάτων. Έχουμε 11 θέματα για διασυνοριακά και διακρατικά προγράμματα και τα προγράμματα από τα 11 αυτά θέματα μπορούν να επιλέξουν 4. Αυτά τα θέματα έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική το 2020 και αυτό είναι καλό. Αλλά το θέμα είναι τι θα συμβεί αν δεν επιλεγούν καθόλου ορισμένα από τα θέματα του καταλόγου αυτού των 11 θεμάτων. Θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινίσουμε αυτή τη θεματολογία και πώς ε, θα εφαρμοστούν τα θέματα αυτά εμπράκτος. Ένα άλλο ζήτημα προκύπτει με τις μακροπεριφέρειες και τη μακροστρατηγική ο σαφής ρόλος των... Ο συγκεκριμένος ρόλος των μακροπεριοχών είναι κάπως ασαφής ακόμη. Λέμε ότι τα προγράμματα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη μακροστρατηγική. Το θέμα είναι ότι οι περιοχές των προγραμμάτων και οι μακροστρατηγικές δεν ε, συμπίπτουν ταυτό ε, πάντα. Τι γίνεται λοιπόν με τη χρηματοδότηση των μακροπεριφερειών. Ο κανονισμός ε, το προβλέπει, αλλά η γνώμη μου είναι ότι δεν θα πρέπει να προβλέψουμε ξεχωριστό προπολογισμό ή επιπλέον κανονισμό για τις μακροπεριφέρειες. Πάντως ο κανονισμός το ρυθμίζει αυτό με ακρίβεια. Αλλά σίγουρα θα γίνουν συζητήσεις και κάποιες ε, διευκρινήσεις θα χρειαστούν εδώ. Τέλος, έχω ένα σχόλιο για τα προγράμματα ENI και ERDI. Νομίζω ότι η διασύνδεσή τους με το μέσο ευρωπαϊκής γειτονίας είναι κάπως ασαφής. Βέβαια, το συζητήσαμε αυτό το θέμα και προηγουμένως και με την Πολωνική Προεδρία, αλλά σίγουρα θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το σημείο, πώς θα σημειώσουμε πρόοδο σε αυτά τα θέματα της γειτονίας για το συνδυασμό των προγραμμάτων με την πολιτική γειτονία. Πάντως, ε, ο κανονισμός ε, έχει πολλά σημαντικά, ε, περιέχει σημαντική πρόοδο για τα θέματα αυτά. Αυτά προς το παρόν από μένα. Περιμένω τα σχόλιά σας και τη συζήτηση. Γιατί η διασυνοριακή συνεργασία είναι σημαντική και σχετίζεται άρρηκτα και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Έχουμε κι άλλους ε, να μιλήσουν ως εισηγητές, αλλά τρία άτομα. Σημαντικό ήταν βεβαίω το τωρινό μας θέμα. Εξίσου σημαντικό βεβαίω είναι και το θέμα της ε, δικής μου έκθεσης ε, δηλαδή τροποποίηση του φυστάμενου κανονισμού. Και μιλάμε βεβαίω για τις ε, έξι εκθέσεις για την... Ε, Έχουμε λοιπόν ε, ένα χαρακτηριστικό που το διαχωρίζει από τις υπόλοιπες πέντε εκθέσεις Δηλαδή δεν αντικαθίσταται εδώ πέρα ένα υφιστάμενος κανονισμός, αλλά έχουμε μια νέα πρόταση κανονισμού, ε, μια επέκταση, μια τροποποίηση και μια βελτίωση σε πολλά σημεία του υφιστάμενου κανονισμού EOS. Ε Ο κανονισμός αυτός λοιπόν υπάρχει από το 2006 δίνει σε τοπικές και περιφερειακές αρχές να κάνουν έναν διασυνοριακό όμιλο εδαφικής ε, συνεργασίας ε, μεταξύ κρατών μελών για με σκοπό ακριβώς να προωθηθεί αυτή η συνεργασία και να μειωθούν οι δυσκολίες όσον αφορά την εδαφική περιφερειακή συνεργασία, επειδή παραδείγματο, χάρη υπάρχουν διαφορετικέ εθνικές διατάξεις και διαδικασία. έτσι, ο κανονισμός αυτός ΕΟΕΣ ε, περιγράφει άρα και ένα νομικό πλαίσιο, δεν ε, σχετίζεται άμεσα και δεν εξαρτάται άμεσα από τα ταμεία, από τα λεφτά, απλά προδιαγράφει ένα πλαίσιο Δηλαδή αυτό υπήρχε ήδη και θα επεκταθεί με τον νέο κανονισμό εντός του οποίου οι υφιστάμενες ε, αυτές ε, πολιτικές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασίας συνεργαζόμενων περιφερειών. Θεωρώ πως στις ερχόμενες εβδομάδες και μήνες ε, θα έχουμε αρκετό χρόνο να δούμε λεπτομερώς την πρόταση κανονισμού και αυτή την πρόταση κανονισμού τώρα κάποιες σοβαρές αλλαγές σε σχέση με τον υφιστάμενο κανονισμό που θα ήθελα να αναφέρω με τη νέα πρόταση κανονισμού η ίδρυση και η αδειοδότηση ΕΟΕΣ διευκολύνεται π.χ. εάν δεν αντιδράσουν εντός εξαμήνου οι εθνικές αρχές τότε θεωρείται πως έχει εγκριθεί ο όμιλος ε, αυτός. Πρέπει λοιπόν ε, να υπάρξει μεγαλύτερη απλοποίηση, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια του δικαίου και βεβαίως ε, θα υπάρχει μια διευκρίνηση των δραστηριοτήτων του ελέγχου. Το δε φάσμα των δραστηριοτήτων για τον Ευρωπαϊκό Ομιλοδαφική Συνεργασία καλύπτει όλες τις πιθανές δραστηριότητες και όχι μόνο όπως μέχρι τώρα την διαχείριση προγραμμάτων και έργων. Άρα οι όμιλοι αυτοί μπορούν να συνεισφέρουν στην εφαρμογή της στρατηγικής ε, για την Ευρώπη 2020 ή μακροπεριφερειακών στρατηγικών και πιστεύω άρα πως συνδέονται στενά με τον κανονισμό για τη διασυνοριακή συνεργασία. Υπάρχει επίσης εδώ πέρα μεγαλύτερη σαφήνεια για τις διαδικασίες προσλήψεων, γιατί βεβαίως ο όμιλος αυτός μπορεί να έχει δικό του προσωπικό και υπάρχει για πρώτη φορά η δυνατότητα ενσωμάτωσης περιφερειών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι ε, πληρώνουμε μία απέτηση διαφόρων μεθοριακών περιοχών που βρίσκονται στα σύνορα ε, με τρίτες χώρες και θα ήθελα να συνεργαστούν. Ε, τώρα ασφαλιστικά ζητήματα για την αστική ευθύνη είναι κάτι το οποίο εμπόδιζε ε, και τυπικά ακόμα την ίδρυση τέτοιων ομίλων ε, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζει νέα πρόταση κανονισμού. Θεωρώ πως ο ΕΟΕΣ ε, θα αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο για να ενισχυθεί η εδαφική συνεργασία, να θεσμοποιηθεί και έχει ήδη από τώρα το πλεονέκτημα πως ο αρχικός κανονισμός του 2006 είχε βεβαίως αποφασιστεί αλλά μέχρι να κυρωθεί από τα κράτη-μέλη περάσανε χρόνια και χρόνια και έτσι οι περιφέρειες που ήθελαν να συνεργαστούν στο πλαίσιο αυτό ε, έπρεπε να περιμένουν. Φαίνεται λοιπόν πως έχουμε εδώ πέρα ένα επιτυχημένο μοντέλο γιατί από το 2006 είχαμε 23 τέτοιους ομίλους και άλλοι 21 είναι σε μια φάση προγραμματισμού και αναμένουν τη νέα τροποποιημένη πρόταση κανονισμού και να τεθεί αυτή σε ισχύ. Χτες ε, το συζητήσαμε στην ομάδα εργασίας ε, και είπαμε πως θα πρέπει να υπάρχει μια ίση αντιμετώπιση των ε, σχεδίων κανονισμού και είπα ήδη πως ο κανονισμός ΕΟΕΣ δεν εξαρτάται από τα κονδύλια, δεν είναι άμεσα συνδεδεμένος από αυτά τα οποία θα γίνουν στο πολιετές πλαίσιο το δημοσιονομικό, αντιθέτως δημιουργεί ένα νομικό πλαίσιο. Οπότε, παρακαλώ την Επιτροπή, ε, όταν ε, λέμε πως δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής, ε, αν υπάρχει άρα η δυνατότητα ο κανονισμός αυτός να εγκριθεί νωρίτερα, από τους άλλους πέντε να το κάνουμε γιατί δημιουργείται έτσι μια βάση εργασίας για τις περιφέρειες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο σε αντίθεση με την υφιστάμενη προγραμματική περίοδο, άρα θα έχουν ένα πλέον έκτημα για να μπορέσουν να εργαστούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τσέλερ. Τον έχει η Μαρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσπαθώντας να τηρήσω ε, αυτό που μας είπε η κυρία Χιμπνερ θα προσπαθήσω να είμαι λακωνική. Ε, εγώ έχω τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχουμε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο Πέραν αυτό όμως θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τέσσερα σημεία. Καταρχήν να επισημάνω την ανάγκη να είμαστε συνεπείς με τη στρατηγική του 2020 και με τους πρωταρχικούς στόχους αυτής της στρατηγικής. Γι' αυτό και χρειάζεται μεγαλύτερη ελαστικότητα στην θεματολογική συγκέντρωση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Δεύτερον, στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην πρόθεση ποιοτικών θέσεων απασχόληση με ιδιαίτερη προσοχή στους νέους, στους ε, πιο ευάλωτους στην στο κοινωνικό αποκλεισμό, στον εξυγχρονισμό των ε, διαφόρων υπηρεσιών απασχόλησης και τη μείωση του υψηλού βαθμού εγκατάλειψης της ε, φίτηση στο σχολείο. Επίσης, ε, να εξαλείψουμε την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να πατάξουμε τη διακριτική μεταχείριση εις βάρος κάποιων ε, μειονοτήτων όπως είναι οι Αθήγανοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ελάχιστε ποσοστώσει για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για κάθε κατηγορία περιφερειών. 25% για τι για για τις περιοχέ τη σύγκληση, 40% για τι μεταβατικέ περιοχέ και 52% ε, για τις περιοχές ε, περιφέρειας ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να ε, βελτιωθεί η συμβολή των ταμείων στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής του 2020, χρειάζονται κάποιες ελάχιστες ποσοστώσεις ή μήπω αρκεί η συνέργεια μεταξύ των ταμείων. Αυτό προβληματίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φυσικά θα πρέπει να απλουστευτεί η διαχείριση, να δώσουμε ε, καλύτερη πρόσβαση των ε, οργανισμών τοπική αυτοδιοίκηση και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στα προγράμματα αυτά, να δώσουμε δηλαδή έμφαση στην περιφερειακή διάσταση. Αυτά για να συμβάλλω και εγώ στη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα υπόλοιπα ταμεία. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Πέρες. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Νικόλα Μάρτιν. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσατε να έρθω στην Επιτροπή σας και να συμμετέχω σε αυτές τις πρώτες συζητήσεις για το πακέτο. Επιτρέψτε μου να επανέλθω στα κύρια ζητήματα που τέθηκαν σήμερα το πρωί και να ξεκινήσω ίσως με το περιεχόμενο των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αστικά ζητήματα και να εξηγήσω τι βρίσκεται πίσω από αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση. Νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό καταρχήν είναι να κατανοήσουμε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις που έχουμε στον κανονισμό για το ΕΤΠΑ, για την αηφόρο αστική ανάπτυξη και τα ελάχιστη, την ελάχιστη χρηματοδότηση του 5% ε, ασφαλώς δεν πρέπει να ε, ειδωθούν ως εκπροσωπευτικά του, των συνολικών επενδύσεων που θα δοθούν στις πόλεις. Γνωρίζουμε ότι οι πόλεις αποτελούν το επίκεντρο μεγάλων επενδύσεων από το ΕΤΜΑ και το Ταμείο Συνοχής τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει ένα, ένα ολόκληρο φάσμα θεματικών, ε, καινοτομία, κοινωνικός αποκλεισμός, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλα ποσά επενδύσεων εν τέλει θα χορηγηθούν σε μητροπολιτικές περιοχές ή σε πόλεις. Το επίκεντρο εδώ είναι λίγο διαφορετικό. Θέλουμε να δοθεί ορατότητα και να προάγουμε και να ενθαρρύνουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων των πόλεων. Μια ενοποιημένη, ολοκληρωμένη προσέγγιση και πάντοτε με στόχο την αηφόραστική ανάπτυξη. Ε, το ποσοστό δικαιολογείται από την ανάγκη να δώσουμε ένα σμπρόξιμο, μια όθηση στα κράτη-μέλη να διαλέξουν τις πόλεις όπου είναι λογικό να εφαρμοστεί μια τέτοια προσέγγιση. Ε, δηλαδή να θα χρησιμοποιηθεί ως ένα είδος μοχλού που θα μας εκτινάξει προς το μέλλον κατά κάποιο τρόπο που θα αποδώσει ωφέλη όχι μόνο στις πόλεις αλλά και στις ευρύτερες περιοχές γύρω από τις πόλεις. Πρόκειται για ένα ελάχιστο όριο, δεν είναι ο στόχος. Δεν λέμε ότι μόνο 5% πρέπει να ξοδέψετε και τέρμα, αλλά ε, ένα ποσοστό πάντοτε μας βοηθά να σμπρώξουμε λίγο τη διαδικασία. Πρέπει λοιπόν αυτό να το δείτε ως κάτι που βαδίζει προς την εκπλήρωση του στόχου της ενοποίησης επενδύσεων από διάφορους τομείς και της ε, παραχώρησης, ε, της παραχώρησης του να επιτρέψουμε στις πόλεις ε, να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά για να υλοποιήσουν το σχετικό στόχο. Είναι επίσης ένα είδος πλατφόρμας. Ε, πόλεις που θα προτείνουν τα κράτη-μέλη, πόλεις που συμμετέχουν στην υλοποίηση αυτών των στρατηγικών, οι οποίες στη συνέχεια θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο για την ανταλλαγή πληροφοριών και την προαγωγή των καλών πρακτικών. Έτσι θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει περαιτέρω κίνητρα και να ενθαρρύνει ακόμα περισσότερο αυτή τη διαδικασία. Και υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο στην πρωτοβουλία να υπάρχουν και κάποια μέσα χρηματοδότησης ε, που θα τα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που θα πηγαίνουν σε συγκεκριμένες δράσεις πιλωτικές ή πειραματικές οι οποίες θα τροφοδοτήσουν την όλη διαδικασία. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα δει τις ενδιαφέρουσες ιδέες που θα προκύψουν από τη διαδικασία αυτή και θα τις βοηθήσει να καρποφορήσουν εντάξει τα αποτελέσματά τους στις πόλεις οι οποίες χρησιμοποιούν τη στρατηγική αυτή προσέγγιση για την αηφόρο ανάπτυξη. Είναι λοιπόν ένα πακέτο το οποίο έρχεται να καλύψει ένα κενό που διαπιστώσαμε στην σημερινή περίοδο, όπου δεν υπάρχει αρκετή ορατότητα των πρωτοβουλειών που λαμβάνονται για τις πόλεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι έτσι θα πληρωθεί αυτό το κενό. δύο-τρία στοιχεία ακόμα για τον κανονισμό για το ΕΤΠΑ. Νομίζω να μιλήσω για τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της χρηματοδότησης για τους συγκεκριμένους ε, κανονισμούς και τις κοινέ διατάξεις. Για παράδειγμα, το βλέπουμε ξεκάθαρα στον τρόπο που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ε, επενδύσεις που να συμβάλλουν στις προτεραιότητες για το 2020. Έχουμε τις 11 θεματικούς στόχους στο γενικό πλαίσιο και μετά έχουμε συγκεκριμένη κείμενα για τη χρηματοδότηση από τα ταμεία για συγκεκριμένα προγράμματα. Γιατί ακριβώς στα, με τα ταμεία είναι που μπορούμε να έχουμε εξατομικευμένες ε, πρωτοβουλίες και εφαρμογές για το πώς θα έπρεπε να συμμετέχουν τα κοινωνικά ταμεία. Φυσικά πρέπει κανείς να το δει συνολικά για να καταλάβει ποιο είναι το νήμα της σκέψης που βρίσκεται πίσω από τα κείμενα. Αυτό ισχύει και για τους δείκτες. Έχουμε δείκτες που είναι ειδικοί για κάθε ταμείο. Ε, γιατί ε, έχει νόημα να έχουμε συγκεκριμένους δείκτες εξατομικευμένους για την προσέγγιση που ισχύει για κάθε ταμείο. Ε, έτσι μπορούμε και να τονίσουμε και να απλοποιήσουμε τη διαδικασία. Θα μπορούμε να παρακολουθούμε καλύτερα τα πράγματα και να αξιολογούμε τι επιτυγχάνεται με τα ταμεία. Και έτσι θα έχουμε μια πολιτική που θα είναι πιο εστιασμένη στα αποτελέσματα και μια πολιτική η οποία είναι streamlined. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν μια σειρά δικτών που είναι υποχρεωτικής εφαρμογής και ε, για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα απλό σύστημα που μας επιτρέπει όμως να αθροίσουμε τα αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δούμε τι γίνεται με τα ταμεία, τι αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί και ποια είναι τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί. Είναι μια επιχειρησιακή, λειτουργική προσέγγιση. Δεν είναι κάτι που το σκεφτήκαμε έτσι ε, χωρίς να το μελετήσουμε, αλλά είναι κάτι που προέκυψε από την κοινή εμπειρία με βάση του δικτύου αξιολόγησης που έχουμε με τα κράτη-μέλη στη συνέχεια για τον ε, κατάλογο των εξαιρέσεων. Υπάρχουν κάποιοι τύποι επενδύσεων που εξαιρούνται. Υπάρχει λοιπόν ένα άρθρο στον κανονισμό για το ΕΤΠΑ, ο οποίος καθορίζει το πεδίο εφαρμογής, αλλά έχει και έναν, αρνητικό κατάλογο για τους πυρηνικού αντιδραστήρες, παραδείγματος χάρη, που, που είναι παντού. Ο λόγος που αναφέρεται η βιομηχανία του καπνού είναι για να είμαστε συνεκτικοί στην προσέγγιση μας. Και θα ήμασταν ασυνεπεί αν λέγαμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ποσά αυτά για να τονώσετε το, τον τομέα του καπνού. Τη στιγμή που υπάρχει σαφώς μια ευρωπαϊκή πολιτική υγείας, στο πλαίσιο της οποίας ε, ε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας που προκαλεί ο καπνός. Είναι θέμα συνοκτικότητας με τις άλλες πολιτικές μας το θεωρούμε δικαιολογημένο και γι' αυτό το συμπεριλάβαμε στις προτάσεις μας. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, ε, ξεκαθαρίζουμε ότι η χρηματοδότηση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσουμε τις προβληματικές επιχειρήσεις. Και αυτό ευθυγραμμίζεται με τις ε, πρακτικές που εφαρμόζουμε γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιοι θα είναι οι εταίροι. Άλλο ζωτικό σημείο. Όπως είπα και χθες, ένα από τα στοιχεία που προσπαθούμε να επιτύχουμε με το γενικό κανονισμό στις κοινέ διατάξεις, ε, τις κοινέ αρχές, είναι να ενισχύσουμε την ε, άποψη αυτή της συνεργασίας, της εταιρική σχέσης σε εθνικό επίπεδο. Φυσικά η ιδέα αυτή υπάρχει. Ε, ανέκαθεν τη θεωρούσαμε θεμελιώδη στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας, τα κράτη δηλαδή να προετοιμάζουν, να καταρτίζουν και να υλοποιούν προγράμματα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να το τονώσουμε, το ενισχύσουμε αυτό, να αναδείξουμε τις καλύτερες πρακτικές έτσι ώστε οι καλύτερες αυτές πρακτικές να διαδοθούν και αλλού και να τις αναγνωρίσουν όλα τα κράτη-μέλη. Και ο μηχανισμός ε, είναι ένας κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος θα υιοθετηθεί με μια πράξη κατεξουσιοδότηση. Εμείς θα φροντίσουμε να συμμετάσχουν οι εταίροι στην προετοιμασία της σύμβασης συνεργασίας ε, και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά όχι μόνο και ευρύτερα όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές και οι φορείς τους. Τώρα, η ακριβής μορφή, συγκεκριμένη μορφή συμμετοχής εξαρτάται από το πλαίσιο που εφαρμόζει το κάθε κράτος μέλος. Δεν μπορούμε να γίνουμε, ε, <clears throat> να ρυθμίσουμε τα θέματα αυτά μέχρι την τελευταία τους λεπτομέρεια. Αυτό ε, πρέπει να γίνει στο εθνικό πλαίσιο. Όσο για τον κώδικα δεοντολογίας, θεωρούμε ότι είναι ένας τρόπος να παρέχουμε ισχυρή καθοδήγηση, κατευθυντήριες γραμμές, να, να, να διαφοροποιήσουμε μεταξύ των διαφορετικών φορέων. Άλλο ρόλο θα παίξουν οι περιφερειακές, τοπικές αρχές και άλλο ρόλο θα παίξουν οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Αυτός νομίζουμε ότι είναι ο σωστός τρόπος για να το κάνουμε. Είναι κάτι βέβαια που μένει να το εξετάσουμε, γιατί τα κράτη-μέλη πρέπει να μας εξηγήσουν τι είδους διαδικασίες εφαρμόζουν αυτά για την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών όταν παρουσιάζεται κάποιο νομοθετικό κείμενο, κάποιος κανονισμός, κάποια ρύθμιση. Για την θεματική συγκέντρωση είναι ένα από τα θέματα που ανέκυψαν και κατά τη χθεσινή συζήτηση. Νομίζω ότι εδώ η αφετηρία είναι και νομίζω όλοι το δέχονται αυτό, ότι υπάρχει ανάγκη συγκέντρωσης των πόρων. Είναι σημείο κλειδί για να επιτύχουμε τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο, την καλύτερη επίδοση. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο. Δεύτερο σημείο. Νομίζω ανέκαθεν θεωρούσαμε απαραίτητο να διαφοροποιήσουμε τι κάνουν τα ταμεία. Γιατί το ε, ESF εστιάζει σε τέσσερις θεματικούς στόχους. ΕΤΠΑ εστιάζεται και στους 11 θεματικούς ε, στόχους. Χρειάζεται λοιπόν μια διαφορετική προσέγγιση για τα δύο ταμεία. Η προσέγγιση λοιπόν που επιλέχθηκε για το ΕΤΠΑ μιλά για συγκέντρωση σε επίπεδο θεματικού στόχου, όχι σε, επίπεδο προτεραιότητας επενδύσεων. Η επιλογή αυτών των τριών κύριων θεματικών στόχων εξηγείται με βάση το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και όλοι το παραδέχονται αυτό. Συνδέονται με τους στόχους για το 2020 και στα πορίσματα του Συμβουλίου. Αυτά είναι τα βασικά. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, ασφάλεια, αποδοτική χρήση της ενέργειας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έρευνα και καινοτομία. Αυτοί οι τομείς αναγνωρίστηκαν και από το Συμβούλιο ότι εκπληρώνουν τις ε, ανάγκες ε, της Ατζέντα 2020 για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και ιδίως για τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές και τις περιοχές σε μετάβαση πρέπει να οριστικοποιηθούν τα ποσοστά για τους θεματικούς αυτούς στόχους. Αλλά στο 80% αυτό υπάρχει ευελιξία ως προς το πώς θα διανεμηθεί αυτό. Το 20% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποδοτική χρήση της ενέργειας θεωρείται ως κλειδί για να εκπληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τους στόχους της, ε, τους ενεργειακούς. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή ε, μάλλον τα κράτη-μέλη προσπαθούν να καθορίσουν τις πρακτικές συνέπειες και για την συζήτηση. Ε, σημαντικό είναι να δούμε εάν υπάρχουν στο έδαφος συγκεκριμένες ανομαλίες που μπορούν να διορθωθούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ε, περιφερειών, περιοχών. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε και όχι να διεξάνουμε τη γενική συζήτηση για το αν το ποσοστό αυτό είναι σωστό ή αν πρέπει να επιλέξουμε ένα διαφορετικό ποσοστό. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι κατά πόσο η εφαρμογή του μηχανισμού αυτού μπορεί να επιλύσει, να διορθώσει κάποιες ε, αθέλητες ε, ανομαλίες. Να δούμε λοιπόν τους σχετικούς μηχανισμούς. Είναι ένα συμβιβασμός, αν θέλετε, μεταξύ του να επιτύχουμε τον καλύτερο το δυνατό αντίκτυπο και να έχουμε και ευελιξία. Η συγκέντρωση Μειώνει βέβαια την ε, ε, ευελιξία, αλλά όχι με τρόπο που να έχει αρνητικές συνέπειες. Εμείς νομίζουμε ότι η ισορροπία είναι η σωστή, γιατί όπως δείχνουν τα στοιχεία υπάρχει ευξημένη πιθανότητα να υπάρχουν τέτοιες ανομαλίες και καλό είναι να τις διορθώσουμε. Και δύο λόγια για το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθούμε να προσφέρουμε κάποιες διατάξεις για τη διασύνδεση μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών, για τη διασύνδεση της πολιτικής συνοχής και της διασύνδεσης της Ευρώπης. Έχουμε συμπεριλάβει λοιπόν κάποιες διατάξεις ως προς το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πολύ σημαντικό είναι στις παράλληλες συζητήσεις για τους δύο κανονισμούς, δηλαδή πολιτική συνοχής και μέσο συνδέοντα την Ευρώπη, σημαντικό είναι να βρούμε έναν συνεκτικό μηχανισμό σύνδεση των δύο. Αυτό που προβλέπεται είναι να υπάρχει ευελιξία. έτσι ώστε η ύψιστη προτεραιότητα να δοθούν σε προγράμματα από τις χώρες συνοχής για τα 10 εκατομμύρια. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν επαρκής ευελιξία για την επίτευξη των στόχων του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη, επιλέγοντας τα πιο σημαντικά προγράμματα και τα προγράμματα που είναι εφικτά. καθώς οι συζητήσεις ε, για το μέσο διασύνδεσης της Ευρώπης, ε, το Connecting Europe Facility, προχωρούν, θα δούμε πώς ε, με τον πιο λογικό και πρακτικό τρόπο θα συνδέσουμε τα δύο. Η βασική ιδέα είναι ότι αυτά τα ποσά χρηματοδότησης θα πάνε στις βασικές υποδομές υπό την άμεση διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη διαβεβαίωση ότι θα ολοκληρωθούν. Αλλά βέβαια θα πρέπει να δούμε τι είναι συμβατό και στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα μεγάλα ευρωπαϊκά έργα που θα εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής. Πρακτικά λοιπόν θέλουμε τα κράτη-μέλη να διαπιστώσουν στο πλαίσιο των μεγάλων έργων υποδομής ποια μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το μέσο διασυνδέοντας την Ευρώπη και ποια, ε, στο πλαίσιο αυτών των μεγάλων έργων ε, της πολιτικής συνογής. Έτσι σκοπεύουμε να προχωρήσουμε. Το Ταμείο Συνοχής και η αποδοτική χρήση της ενέργειας στον τομέα των νοικοκυριών. Ε, αυτό είναι ελαφρώς διαφορετικό ζήτημα. Το, πολιτικό, το Ταμείο Συνοχής έχει τη δική του λογική και εστιάζεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα, στην περιβαλλοντική υποδομή και θεωρούμε καλό να διατηρηθεί αυτή η προσέγγιση. Τώρα, η αποδοτική χρήση της ενέργειας στα νοικοκυριά εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ΕΤΠΑ. Εμείς το βλέπουμε έτσι, γιατί έτσι επιτυγχάνεται μια καλή ισορροπία στη χρήση των ταμείων, των πόρων των ταμείων. Κατανοώ ότι για μερικά κράτη-μέλη αυτό μπορεί να αποτελεί και πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα με, να ανοίξουμε το Ταμείο Συνοχής ε, είναι να χάσουμε αυτή την επικέντρωση. Ε, και να δώσουμε τους πόρους του Ταμείου Συνοχής σε τομείς για τους οποίους δεν προορίζονταν. Και λίγα σχόλια τώρα για τον κανονισμό για το ETC, για την εδαφική συνεργασία προβλέπεται αύξηση της χρηματοδότησης, γιατί αναγνωρίζεται η μοναδική σημασία της εδαφικής συνεργασίας και το γενικό πλαίσιο της ε, πολιτικής συνοχής. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα να έχουμε έναν ξεχωριστό κανονισμό για την εδαφική συνεργασία σε αναγνώριση της σημασίας της και για τη διευκόλυνση επίσης ε, της υιοθέτηση ενός σαφούς πλαισίου. Γι' αυτό έχουμε εισαγάγει διάφορα στοιχεία Κάτι άλλο σημαντικό είναι να ενισχυθεί η διασύνδεση μεταξύ της εδαφικής συνεργασίας και μεγάλων προγραμμάτων, μεγάλων έργων. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τις ε, συμφωνίες συνεργασίας, όπου γίνεται και αναφορά στις προτεραιότητες. Έτσι δίνουμε κίνητρα στο κράτος μέλος, ε, στα κράτη-μέλη, δείχνοντάς τους ότι έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση. Τώρα για τις στρατηγικές. Θέλουμε να ενισχύσουμε και την μακροπεριφερειακή στρατηγική. Εν μέρη αυτό γίνεται με τους ε, συμβάσεις συνεργασίας, όπου τα κράτη-μέλη θα καθορίσουν οι ιεραρχίες, μια ιεράρχηση των στρατηγικών τους και θα αναφέρουν τι θα κάνουν για την μακροπεριφερειακή στρατηγική, αλλά και στον κανονισμό για την εδαφική συνεργασία. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες επενδύσεων οι οποίες θα επιτρέψουν χρηματοδότηση από τα διακρατικά προγράμματα για την μακροπεριφερειακή στρατηγική. Και, αυτός είναι ένας πολύ, και αυτή είναι μια πολύ συγκεκριμένη, ένα πολύ συγκεκριμένος τρόπος διασύνδεσης. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι τα κάλυψα τα κυριότερα. Ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you, very much indeed for your details. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις δηλώσεις σας και τις απαντήσεις σας. Τώρα έχει φτάσει η ώρα να δώσουμε το λόγο στους ε, βουλευτές. Ε, σύμφωνα με τον κατάλογό μου, ο κύριος Ντέαντζελης είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, εν συντομία, ε, για τον κανονισμό για την εδαφική συνεργασία. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο κατά τη γνώμη μου. Κυρίως για την ανάπτυξη, για την οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση. Ένας πρώτος στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας, κατά τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι ο κανονισμός πρέπει να επιδιώξει το στόχο στήριξης της μέγιστης δυνατής συνεργασίας μεταξύ των χωρών. Ακριβώς επειδή η, συνεργασία, η εδαφική συνεργασία πολύ συχνά βοηθά στην επίλυση προβλημάτων μιας χώρας ή μιας περιφέρειας ή μιας περιοχής, τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν ε, μέσα στα εθνικά ή περιοχικά σύνορα. Και πρέπει πραγματικά να, το ευνοήσουμε αυτό, να ευνοήσουμε την, ε, ε, τη διάδοση των καλών πρακτικών να βελτιώσουμε τους τομείς, τις επενδύσεις, τις δράσεις και αυτό κυρίως μέσω της καλής χρήσης αυτών των πόρων. Να στηρίξουμε και να ευνοήσουμε τους στόχους της ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό στον νέο προγραμματισμό να επιτευχθεί μια πιο συγκεκριμένη συμφωνίας, πιο συγκεκριμένης για τα χρηματοδότηση έργα. Και αυτό μέσω, της, ε, μέσω πολύ σαφών στόχων. Όταν οι στόχοι είναι σαφείς ε, και καλά καθορισμένοι, όλα πάνε καλά. Τα προγράμματα πρέπει να αντιστοιχούν στις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρώπης. Πρέπει να συνδεθούν λοιπόν με τις στρατηγικές που προτείνουν τόσο τα κράτη-μέλη όσο και οι περιφέρειες. Και όλο αυτό στο πλαίσιο ενός πολύ καλού συντονισμού. Περισσότερος συντονισμός, περισσότερη ενοποίηση και ολοκλήρωση μεταξύ εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων. Και έρχομαι στο τέλος της παρέμβασής μου. Ένα σημείο που μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό είναι η απλοποίηση. Να... Απλοποιώ σημαίνει επιταχύνω. Επιταχύνω σημαίνει <clears throat> προχωράω. Αυτό είναι ο πιο σημαντικός στόχος. Μέσω της μείωσης των ε, γραφειοκρατικών και διοικητικών βαρών στην ε, διαχείριση των προγραμμάτων. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μια δημόσια διοίκηση κατά τη χρήση αυτών των πόρων που να είναι φιλική. Φιλική προς τις επιχειρήσεις, φιλική προς τους πολίτες. Γι αυτό και ε, σε αυτό συντείνει ο στόχος της απλοποίησης. Εν για τις δαπάνες. Πέρα από το ύψος των επενδύσεων, θα συζητήσουμε για τους αριθμούς, αλλά πολύ σημαντική είναι η ποιότητα της δαπάνης και η καλή χρήση, η χρηστή χρήση αυτών των πόρων. Οι πόροι πρέπει να πάνε σε προγράμματα ε, ποιοτικά. Και αυτό θα καταστεί δυνατό μόνο αν ε, <clears throat> επεξεργαστούμε κανόνες που να διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ, Φραντσέσκο. Θα αναπληρώσω λίγο την κυρία Χίμπνερ και θα κλείσουμε τώρα τον κατάλογο των ομιλητών. Έχουμε νέοι ομιλητές και 20 λεπτά ακόμα. Οπότε να σας παρακαλέσω να περιοριστείτε σε δύο λεπτάκια ο καθένας και τώρα ε, είμαι εγώ η επόμενη ομιλήτρια. Τέλος πάντων, δεν είναι πολύ δίκαιο, οπότε ακούσουμε τώρα την κυρία Ένστ. Α, γρήγορα ήρθε η σειρά μου. Θα ήθελα ως κοιόδης εισηγήτρια για την ομάδα μας να πω κάποια πράγματα. Ξανά για την ε, θεματική αυτή συγκέντρωση. Δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με αυτά τα οποία μας είπε εδώ πέρα ο κύριος Μάρτιν. Γιατί δείτε εδώ πέρα παραδείγματος χάρη τις ανεπτυγμένες και τις ε, μεταβατικές περιοχές όπου 80% ε, των ε, ποσών του ΕΤΠΑ θα χρησιμοποιηθούν στα άρθρα 1, 2, 3 και μετά έχουμε το 20% γιατί μένουν κάποιες, κάποιοι τομείς εκτός ή δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία δεν είναι σαφές ή υπάρχουν θεματικοί στόχοι ή δεν υπάρχουν είναι ούτως ή άλλως περιορισμένοι δεν χρειάζεται να τους περιορίζουμε κι άλλο ε, εξάλλου αφαιρείται εδώ πέρα ευελιξία. Έχουμε πολύ διαφορετικές περιοχές. Έχουμε τόσο διαφορετικές περιοχές στη Γερμανία. Όχι μόνο όσον αφορά το ΑΕΠ, αλλά όσον αφορά τη συνολική τους ανάπτυξη. Και έτσι πιστεύω πως η, ε, ο περαιτέρω περιορισμός ε, δεν είναι θετικός. Γιατί πρέπει να είναι έτσι οπωσδήποτε τα πράγματα. Επίσης, κάτι άλλο έχω πρόβλημα. Αν δείτε τους κοινούς δείκτες που λένε περιβάλλον και κλίμα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη σημασία, ε, δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη με τις συγκοινωνίες, γιατί υπάρχει εδώ πέρα μόνο ποσοτική, ποσοτικός ορισμός, δεν υπάρχει κανένας ποιοτικός ορισμός. Ε, τώρα δεν θέλω να τα κάνουμε όλα μέχρι τις λεπτομέρειες, αλλά λέτε εδώ πέρα νέους δρόμους. Ε, δεν ε, <coughs> επαρκούν αυτά νομίζω για να επιτύχουν και τι άλλο, τι άλλο αστική διάταξη ναι ευχαριστώ για τη δήλωσή σας ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν ξέραμε τι εννοούμε εδώ πέρα αλλά τίθεται το ζήτημα το εάν ε, αρκεί αυτό θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις σας ευχαριστώ Εάν και οι άλλοι ομιλητές περιοριστούν σε τόσο χρόνο θα ήταν υπέροχα τα πράγματα. Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Ένα, ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι θα μιλήσω. Κοιτάξτε, δύο μηνύματα έχουμε τώρα πρώτα απ' όλα. Για την ε, δαφική συνεργασία, πράγματι δικαίως το συνδέουμε με τα εξωτερικά σύνορα, πολιτική γειτονίας, και ε, το είπε αυτό και η Επιτροπή Εξωτερικών νομίζω στην έκθεση που είχε ψηφιστεί πρόσφατα που έκανε δεκτή την ε, πρότασή μας στη γνωμοδότηση της κυρίας Μπομπίνσκα νομίζω ήταν αυτό ότι θα πρέπει να αποτελέσει αυτό βασικό αντικείμενό μας όσον αφορά και τη χρηματοδοτική πτυχή αλλά και την διαχείριση των προγραμμάτων αυτών στο πλαίσιο της πολιτικής ε, γειτονίας. Ε, υπάρχει λοιπόν, ε, από ό,τι κατάλαβα, μια θετική αντιμετώπιση στην Επιτροπή Εξωτερικών. Είτε μιλάμε για τη γενικότερη γειτονία μας, είτε όντως πραγματικά για τις μεθοριακές περιοχές και την προσέγγιση που έχουμε εκεί για μια ανάπτυξη. δεύτερη παρατήρηση, πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα είναι η θέση της σύμβασης αυτής της εταιρικής σχέσης ε, και από αυτά τα οποία μας είπατε αντιλαμβάνομαι πως έχει κατά κύριο λόγο να κάνει με τους εταίρους εντός των κρατών μελών και εάν ε, γίνει αυτό σωστά δεν θα μπούμε στη συζήτηση περί μακροαιρεσιμότητας καθώς βεβαίως αυτό έχει συνδεθεί με εντάσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά μπορούμε να τα αφήσουμε νομίζω εκτός. Για να συζητήσουμε πραγματικά περί ε, πολιτικής ε, γιατί δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε με σε επίπεδο κρατών μελών ε, και εμείς θέλουμε νομίζω να πούμε πως όσο μεγαλύτερη θα είναι η συνεκτικότητα τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επιτυχία. Μάλιστα ευχαριστώ η κυρία Ραμάνο Μανέσκου. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση Olbricht και κατόπιν να σχολιάσω αυτά που είπε ο κύριος Μάρτιν. Εγώ ουδέποτε δεν αμφισβήτησα τις αγαθές προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά το σχέδιο εμ, ανάπτυξης των πόλεων και τον κατάλογο με τις 20 πόλεις. Αυτό που είπα είναι ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, ώστε τα σχέδια αυτά που γενικώ είναι ποιοτικά γιατί προωθούν την ανάπτυξη, να φροντίσουμε ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στις τοπικές ανάγκες, στην τοπική πραγματικότητα. Δεν αρκούν εδώ οι αγαθές προθέσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να ελέγξουμε με ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή αυτών των 20 πόλεων και το ποσοστό του 5% ίσως δεν είναι η καλύτερη μέθοδος. Καλό θα ήταν να έχουμε ένα κατάλογο αστικών ζωνών και όχι μόνο έναν περιορισμένο κατάλογο 20 πόλεων. Θα πρέπει να διαβρύνουμε κάπως τη σφαίρα. Τώρα σε μια άλλη πτυχή Αναφέρθηκε ότι μια εταιρεία που έχει πάνω από 50, απασχολεί πάνω από 50 εργαζομένους δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κοινοτικά κονδύλια για στόχους πλήν έρευνα και τεχνολογικής ανάπτυξης. Και πάλι θα πρέπει να είμαστε γεωμένοι. γιατί για να έχουμε ισότιμη πρόσβαση και των μικρομεσαίων και των, των μεγάλων επιχειρήσεων στα κονδύλια, πιστεύω ότι όλοι θα βγουν κερδισμένοι. Στο σημείο αυτό λοιπόν περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία πρόταση που θα ανταποκρίνεται πιο πιστά στην πραγματικότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ταμείο Συνοχής. Έχουμε πρόβλημα με αυτή την μακροαιρεσιμότητα. Γιατί φαίνεται να μην υπάρχει ε, σχέση μεταξύ τη, της πολιτικής ε, ε, ανάπτυξης, εδαφικής ανάπτυξης μιας χώρας και το, το κονδυλίων που λαμβάνει. Επίσης, τι θα γίνει με τη χρηματοδοτική διευκόλυνση, αυτό το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Η, είδαμε ότι σημαντικά κονδύλια θα μεταφερθούν από το Ταμείο Συνοχή σε αυτό το μέσο διευκόλυνση. Το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια ε, αυτά τα κράτη-μέλη για να χρηματοδοτήσουν ορισμένα σχέδια. Πρέπει να είναι τα βέλτιστα σχέδια. Θέλουμε τα καλύτερα προγράμματα και να δούμε ε, πώς θα χρησιμοποιήσει κάθε χώρα το μέσο αυτό διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριο Σαλφόνση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω για την εδαφική συνεργασία και ένα πολύ ανησυχητικό θέμα τα θαλάσσια σύνορα. Ε, η συνεργασία στο επίπεδο ΝΑΤΣ 3, όταν έχουμε νησιά όπως η Κορσική και η Σαρδινία, δεν μπορούμε δαφική συνεργασία να την περιορίσουμε στο βόρεια Σαρδινία και την νότια Κορσική. Έχουμε ένα περιορισμό που είναι παράλογος κατά τη γνώμη μας. Και για το όριο των 150 χιλιόμετρων θα μπορούσαμε να έχουμε συνεργασία με τις Βαλεαρίδες νήσους ή συνεργασία για την τουριστική ανάπτυξη, γιατί σίγουρα έχουμε πολλά κοινά σημεία. Οι Βαλεαρίδες βέβαια απέχουν πάνω από 150 χιλιόμετρα από την Κορσική, άρα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με βάση τον όρο, τον περιορισμό αυτό. Έχουμε μια υπηρετική προσέγγιση που δυστυχώς ε, αδιαφορεί για τις ε, θα, νησιωτικές περιοχές. Αντίθετα, στα νησιά θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε ε, προγράμματα συνεργασίας μεταξύ Βαλένσιας και Ιταλίας για να χρησιμοποιήσουμε και τη θαλάσσια δίωδο. Αλλά δυστυχώς εξαιτία του περιοριστικού χαρακτήρα αυτού του κανονισμού ΝΑΤΣ 3, 150 χιλιόμετρα, αποκλείονται αυτά τα προγράμματα. Θέλουμε εξαίρεση τουλάχιστον για τις νησιωτικές περιοχές και για προγράμματα που, ξε, που ξεπερνάνε θαλάσσια σύνορα, γιατί μιλούμε για προγράμματα που έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μακροπεριφέρειες, ε, με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσθέτει αυτό το όργανο στη, στην παρακολούθηση της εδαφικής πολιτικής και σίγουρα οι μακροπεριφέρειες ε, έχουν προβλήματα σε ορισμένες περιοχές εξαιτίας των σύνορων και μερικές είναι πιο περιορισμένες από άλλες Χρειαζόμαστε όμως μια συνολική προσέγγιση, μια συνέπεια και να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτή την μακροπεριφερειακή στρατηγική. Ευχαριστώ. Η κυρία Γουκατσέφσκα. Σας ευχαριστώ. Εγώ έχω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το θέμα του αποκλεισμού της στήριξης συγκεκριμένων προγραμμάτων εγώ κατάγομαι από μια περιοχή που είναι καπνοπαραγωγός και άκουσα ότι ο αποκλεισμό αυτός, ε, όπως είπε ο κύριος Μάρτιν, ε, δικαιολογείται ε, από τις προτεραιότητες μας στην πολιτική υγεία στον καταναλωτό. Θέλουμε να περιορίσουμε την καπνοπαραγωγή. Τότε τέτοιος αποκλεισμό δεν θα πρέπει να ισχύει μόνο για το καπνό, θα πρέπει να συμπεριληφθεί ε, και να συμπεριληφθούν και τα πνευματόδι ποτά, η παραγωγή τροφίμων fast food. Δεν με πείθει το επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η πολιτική υγεία των καταναλωτών συνέβαλε στον αποκλεισμό μόνο και μόνο του καπνού της καπνοπαραγωγής από τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Γνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Κοινωνικό Ταμείο σε ό,τι αφορά την αύξηση του επίπεδου απασχόλησης, κυρίως για, για τον περιορισμό της ανεργίας των νέων. Δυστυχώς οι νέοι είναι αυτοί που περισσότερο μαστίζονται από την ανεργία και πολύ συχνά βλέπουμε κάποιες γενικές παρατηρήσεις για την ενεργό ένταξη, για παράδειγμα το θέμα κοινωνικής ένταξης ή ε, συμπερίληψη των, ε, μειονοτικών, των μειονοτήτων που είναι πιο ευάλωτοι στον αποκλεισμό. Αναφέρονται εδώ οι Αθήγανοι. Γιατί περιοριζόμαστε στους Αθήγανους, γιατί δεν αναφερόμαστε στους μετανάστες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε πάγια μέσα ή στην ε, αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Όταν μιλούμε για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, γνωρίζουμε ότι οι ποιοτικέ ε, υγειονομικέ υπηρεσίες θα είναι και δαπανηρέ, δεν θα είναι καθόλου φθηνέ. Παρόμοιες παρατηρήσει έχω πολλές και διάφορες. Η ισότητα των δύο φύλων. Γιατί εδώ δεν περιλάβαμε και μια διάταξη για την εξάλληψη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών, που είναι μια έκφραση τη ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Το θέμα τη ε, μισθολογική ανισότητα το επισημαίνουμε πολλέ φορέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ένα γενικό θέμα, η αποτελεσματικότητα τη ε, χρήση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακή Ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία χώρα ε, που ε, δεν κατάφερε να χρησιμοποιήσει κοινοτικά κονδύλια για επαναφορά στην αγορά των ανέργων. Ή δεν λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα επαγγέλματα, συγκεκριμένε ε, δεξιότητε. Νομίζω ότι εκεί θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια και εκεί να φανεί η αποτελεσματικότητά του. Αυτό είναι σημαντικό και για τι στατιστικέ. Δυστυχώ δεν υπάρχουν τέτοια στατιστικά στοιχεία για την αποτελεσματική χρήση των κοινωτικών κονδύλιων. Τέτοιου είδους παρατηρήσεις ε, για καταρτήσεις που διευκολύνουν την επαναφορά στην αγορά νομίζω είναι και καλός μετρήσιμος δείκτης για το πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιούνται τα κονδύλια. Κύριε Στρεμόπουλος. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να τονίσω και εγώ για αυτό τον ε, κανονισμό, τον 1084 κάθετος 2006, ότι είναι ένας ε, μικρός, ε, νέος και μικρός σχετικά κανονισμός και πράγματι έχει αρκετές βελτιώσεις. Η Επιτροπή έχει προτείνει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται και εκτελείται η πολιτική για τη συνοχή. Σημεία όμως, όπως η συγκέντρωση της χρηματοδότησης σε ένα μικρότερο αριθμό προτεραιοτήτων που συνδέονται περισσότερο με τη στρατηγική της Ευρώπης του 2020, η επικέντρωση στα αποτελέσματα, η παρακολούθηση της προόδου ε, προς την επίτευξη των ε, συγκεκριμένων και συμφωνημένων στόχων, ε, η απλούστευση των διαδικασιών, συγκαταλέγονται πραγματικά στα σημαντικά στοιχεία αυτής της πρότασης. Τα σημεία που εμείς ως πράσινοι δίνουμε βαρύτητα είναι, ως γνωστόν, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ενεργειακή αποδοτικότητα και οι ενενιώσιμες πηγές ενέργειας, η επέκταση των χρηματοδοτικών ευκαιριών για την κλιματική αλλαγή, αλλά σημαντικότερο όλων για μας είναι η πρόληψη των κινδύνων. Και εδώ μέσα έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι είναι πολύ καλύτερο να προλαμβάνεις από το να πληρώνεις αφού συμβεί το κακό. Μάλιστα κάποιος ε, από την Κομισιόνα. Ο ομιλητή, είχε πει, ε, είχε κάνει λόγο για 7 προ 1. Ο λόγος, ε, ε, λοιπόν, για έναν παραπάνω λόγο, μπορούμε να έχουμε τη βέλτιστη αποδοτικότητα αν αξιοποιούμε τα κονδύλια στην πρόληψη παρά στην εκ των αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών. Επιπλέον, η απευθεία σύνδεση με τις οδηγίες για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών που συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό, οι θαλάσσιες υποδομές σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο η προστασία της βιοπικιλότητας είναι όλα σημεία που εντοπίσαμε σε αυτόν τον κανονισμό. Ένα σημείο που θα ήθελα να προτείνω είναι να προσθεθούν στον κανονισμό οι δυνατότητες χρηματοδότησης για τις περιοχές Natura 2000 που τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλές άλλες δεν έχουν ενισχυθεί επαρχώς ανάμεσα σε άλλα και με χρηματοδοτικά εργαλεία. Σας ευχαριστώ πολύ. So, vielen Dank. Ähm, Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα είμαι εγώ η τελευταία ομιλήτρια πριν από τον εισηγητή και θέλω να τονίσω ότι εκπροσωπώ την κυρία Βέσφαν η οποία είναι στην αίθουσα αλλά δεν μπορεί να μιλήσει, μπορεί μόνο να ακούσει. Είναι σκιοδησηγήτρια για το ΕΤΠΑ, για την ομάδα μας και μου πρέπει να πω κάποια πράγματα. Η ομάδα συμφωνεί πλήρως με την ε, πρόταση της ε, Κομισιόν πως πρέπει το ε, ΕΣΠΑ το, να περιοριστεί σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα και να μην κάνουμε τα πάντα χωρίς κάποια αποτελεσματικότητα. Και βεβαίως θα πρέπει μία περιοχή η οποία ε, πλήττεται από δημογραφικές εξελίξεις, ε, έχει διαφορετικές προτεραιότητες από μια άλλη η οποία δεν ε, έχει κάτι τέτοιο. Οπότε θα πρέπει να δούμε λεπτομερώς εάν οι στόχοι που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά μπορούν να προωθηθούν ή μήπως οδηγούμαστε σε μένες εξελίξεις. Αυτό το οποίο λοιπόν είναι ιδιαίτερο δύσκολο είναι οι περιοχές οι οποίες είναι καλύτερα ανεπτυγμένες να μην κάνουν πλέον διαρθρωτικά μέτρα. Θεωρώ πως ε, υπάρχει εν μέρει ανάγκη και σε αυτές τις περιοχές και πλήρης απαγόρευση τέτοιων ε, μέτρων δεν ε, ανταποκρίνεται νομίζω στα αλήθεια στις προτεραιότητές μας. Όσον αφορά τώρα την αστική ανάπτυξη υπάρχουν κάποια ερωτηματικά που δεν απαντήθηκαν βεβαίως όλα. Θα σας πω 20 πόλεις ανακράτος μέλος, εντάξει, για το Λουξεμβούργο μπορεί να ακούγεται καλό ή στη Γερμανία θα έχουμε προβλήματα. Θεωρώ πως η παλιά κοινοτική πρωτοβουλία νομίζω θα πρέπει να αναβιώσει. Την είχαμε καταργήσει γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλο διοικητικό κόστος. Ένα παραδείγματο χάρη σε ένα ομοσπονδιακό κρατήδιο στη Γερμανία μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μόνο μία πόλη και πάλι αυτό να το κάνει το κράτος μέλος και όχι οι περιφέρειες. Ε, εδώ πέρα έχουμε ξεφύγει τελείω από την προσέγγιση της περιφερειακής πλέον πολιτικής. Οπότε αν πούμε η απόφαση είναι των κρατών μελών και ε, δεν μπορεί να γίνει ποτέ, αλλά τότε νομίζω πως είναι λανθασμένη η απόφαση. Συνολικά λοιπόν χρειάζεται περισσότερη ευελιξία στον κανονισμό που μπορεί να συμβαστεί βέβαια με τις προτεραιότητες, αλλά νομίζω πως θα έχουμε έτσι την ευκαιρία να συνεργαστούμε στενά με τον ε, κύριο εισηγητή. Αυτά από την κυρία Βέστφαλν τώρα. Να δώσω τον λόγο ξανά στη Μαρία, την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι επιγραμματική. Μετά τι παρατηρήσει του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι δεν χρειαζόμαστε επιλεκτική μνήμη εδώ και η σημαντική οικονομική και κοινωνική σύγκληση που επέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν θα πρέπει να λησμονείται. Αλλά φυσικά στη διαχείρισή μα ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα. Η περιφερειακή πολιτική δεν περιορίζεται σε ορισμένου μόνο Θα πρέπει να καταργηθεί η μακροοικονομική αιρεσιμότητα γιατί η αιρεσιμότητα αυτή ε, δεν θα πρέπει να συνδυάζεται με κυρώσει της πολιτικής ε, συνοχής, γιατί αυτό, αυτό θα είναι διπλή κύρωση. αφαίρεση του κονδυλίου και αδυναμία α, τήρησης των υποχρεώσεων και φυσικά αποκλεισμό από περαιτέρω κονδύλια. Τρίτον, η, η, το αποθεματικό αποτελεσματικότητας. Ε, αποθεματικό ε, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να στηριζόμαστε σε θετικά αποτελέσματα και όχι σε μεταφορά ε, κονδυλίων προ πιο αποδοτικά προγράμματα. Τέταρτον, έχω πολλέ αμφιβολίε για την εξάντα και εξπόστ αιρεσιμότητα. Και οι δύο μορφέ αιρεσιμότητα είναι υπερβολικέ κατά τη γνώμη μου, με τη μορφή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομα, η κυρία Μάνερ. Ένα λεπτό. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Σύντομα κάποια σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα κύριε, ή τον κύριο Ντεάντζελη, συμφωνώ με αυτά τα οποία είπατε για να ενισχύσουμε αυτό τον κανονισμό πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση και να υπάρξει και συντονισμός με τις άλλες πολιτικές, απλοποίηση πολύ σημαντική καθώς και το ζήτημα της ποιότητας ε, των δαπανών και μείωση της δημόσιας ε, διοίκησης. Μετά για ο Λάμπερτ Φανίστελ Ρόι ανέφερε τη σύνδεση με την ευρωπαϊκή γειτονία και Της, ε, την εδαφική συνεργασία και βεβαίως θα συζητηθεί αυτό το θέμα σε 6 Δεκεμβρίου, θα συνεργαστούμε. Είναι λοιπόν σημαντικό να προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε τα προγράμματα αυτά. π.χ. μπορεί να γίνουν έτσι ευκολότερα τα προγράμματα αυτά εργασίας. Μετά κάποια σχόλια ε, για τον κύριο Αλφονσί. Γνωρίζω την προβληματική συζήτηση περί των 150 μέτρων, της απόστασης δηλαδή, γιατί θέλω να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα για τις μακροπεριφέρειες. Ξέρω πώς κάνετε αυτή την έκθεση και θα ήθελα να συνεργαστούμε για το ζήτημα των μακροπεριφερειών. Είναι πολύ σημαντικό τα ζητήματα αυτά να είναι πιο ξεκάθαρα στον κανονισμό. Και ευχάριστο το ότι ακούσαμε τον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν να λέει πώς μπορεί να υπάρξει πιο στενή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος τον λόγο. Ε, να παρακαλέσω τώρα οι σίτες ε, να αναβάλουν τις ε, υπόλοιπες παρεμβάσεις τους για την επόμενη συνεδρία. Σε ένα λεπτό δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Θα ήθελα όμως να δώσω την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Διευθυντή, τον κύριο Πακέ, της Γενικής Διεύθυνσης ΜΟΥΒ, για να αναφέρει, να απαντήσει σε κάποια ε, ερωτήματα τα οποία ακούστηκαν. Μια στιγμούλα, Γιάν, με συγχωρείτε κυρία Πρόεδρε, εγώ λέω να μείνουμε στο πρόγραμμα που έχουμε. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές ε, που μπορεί να τους ενδιαφέρει αυτό. Το μέσο αυτό είχε προγραμματιστεί για τι ώρα, τώρα. Ε, πριν από μισή ώρα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει, λέει ο πρόεδρος. Μάλιστα, γιατί μπορεί κάποιος βουλευτής να ήθελε να τα ακούσει. Α, εντάξει. Όχι, θα ξεκινήσουμε τη μελέτη στις 11.30 και κανονικά έπρεπε να έχουμε ήδη συζητήσει το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Οπότε οι παρατηρήσεις του εισηγητή την επόμενη φορά. Ο κύριος Πακέ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω το χρηματοδοτικό μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντική η επιτροπή σας, λόγω της συμπληρωματικότητας που χρειάζεται μεταξύ του μέσου αυτού ε, συνδέοντα στην Ευρώπη και των ε, διαφόρων μηχανισμών ε, περιφερειακής πολιτικής. Το μέσο αυτό συνδέεται στην Ευρώπη υιοθετήθηκε πριν από ένα μήνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τμήμα του συνολικού πακέτου προτάσεων που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συμβάλλει στο πρόγραμμα ενίσχυσης οικονομικής ανάπτυξης Ευρώπης, Συμπλήρωση τη ε, εσωτερική αγορά με ε, ακρογωνιού λίθους ε, το, επικοινωνία ενέργεια, μεταφορές, ανταγωνιστικότητα. Το μέσο αυτό ενισχύει τις συνέργειες και δίνει προστιθέμενη αξία. Στόχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να βρεθούν οι κατάλληλες συνέργειες μεταξύ των τριών τομέων Επίσης προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει συνέργειες και καλύτερη ένταξη μεταξύ των πλαισίων πολιτικής και σχεδιασμού που προβλέπονται τις κατευθυντήριες γραμμές για τις, ε, πληροφορι... για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, την ενέργεια και τις μεταφορές, καθώς και τα ευρωπαϊκά μέσα για τη στήριξη αυτής της εφαρμογής. Η χρηματοδοτική διευκόλυνση συνέοντας στην Ευρώπη αποτελεί σημαντικό στοιχείο του συνολικού χρηματοδοτικού πλαισίου, αλλά θα πρέπει να ε, θεωρηθεί και σε συνδυασμό με τις ε, γενικές κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να υποστηριχθεί η βιομηχανία, να υποστηριχθούν τα κράτη-μέλη και να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα διευρωπαϊκά δίκτυα που είναι και ο νοτιός μυαλός της εσωτερικής αγοράς και συμβάλλουν στην συνοχή της ευρωπαϊκής, ε, το, της ευρωπαϊκής επικράτειας. Προσπαθήσαμε ε, να δούμε πού δικαιολογούνται κρατικά κονδύλια για το μέσο αυτό. Ε, υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφόρων σχεδίων και μάλιστα λάβαμε υπόψη αυτό στους τρεις τομείς και στο μέσο αυτό διευκόλυνσης υπάρχουν κάποιες διατάξεις για καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση σχεδίων και όπου διαπιστώσαμε ότι χρειάζονται και δημόσια κονδύλια προχώρησαμε ακόμη περισσότερο, προσπαθώντας να διαπιστώσουμε πού αυτά τα δημόσια κονδύλια θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκά. Και το χρηματοδοτικό μέσο συνδέοντας Ευρώπης φυσικά απαιτεί και κοινοτικά κονδύλια για το ευρωπαϊκό σχέλος των 10 t 10 e και 10 ict το Διευρωπαϊκό Δικτύο Ενέργειας, Μεταφορών και πληροφοριών, Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Προσπαθήσαμε να βρούμε και κάποιες διασυνδέσεις με άλλες πολιτικές και δημοσιονομικά μέσα, για παράδειγμα το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας που θα υποβληθεί αυτή την εβδομάδα. Επίσης σχέση με την εξωτερική διάσταση των τριών τομέων που είναι σημαντική και φυσικά και της περιφερειακής χρηματοδότησης επίσης σημαντική. Το χρηματοδοτικό μέσο συνδέοντας στην Ευρώπη ε, θέλει να είναι συμπληρωματικό, εν μη διάλογο απόλυτα συνεπές και συναφές με, τις, με τα άλλα μέσα της περιφερειακής πολιτικής. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, τα διάφορα εργαλεία των περιφερειακών πολιτικών θα πρέπει να ενισχύουν την ευρυζωνία, ενώ το συνδέοντας στην Ευρώπη θα καλύψει στοιχεία της ευρυζωνίας που δεν είναι περιφερειακά ή δεν, θα, δεν μπορούν να υλοποιηθούν εθνικά. Πάντω, ευελπιστούμε ότι τα κράτη-μέλη θα, θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία τη περιφερειακή πολιτική για διανομή, δίκτυα σε τοπικό επίπεδο, για την ενεργειακή αποδοτικότητα, που είναι σημαντικό στόχο και προτεραιότητα και θα πρέπει να παραμείνει ύψιστη προτεραιότητα, ενώ το μέσο ιδέοντα τη Ευρώπη θα επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό ε, προτεραιοτήτων, προκειμένου να συμπληρώσει την ευρωπαϊκή ενεργειακή διάσταση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, το μέσο ιδέατος στην Ευρώπη σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά, δεν υποκαθιστά ε, τα, τα, το Ταμείο Συνοχής ή τα κονδύλια της συνοχής που επικεντρώνονται στις υποδομές των μεταφορών και στα συστήματα των διευρωπαϊκών δικτύων. Ε, κυρίως αφορούν τα δίκτυα Core Network και Comprehensive Network. Επίσης επικεντρώνεται στα διασυνοριακά στοιχεία των Core Networks και επικεντρώνεται και σε σχέδια που είναι, αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες αυτό το Core Network. Το πλαίσιο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ή προτείνει στα κράτη-μέλη να αναλάβουν δεσμεύσεις ώστε μέχρι το 2030 να παρουσιάσουν ένα ενσωματωμένο core network στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα καλύπτει και τα 27 κράτη-μέλη, ολόκληρη την ενιαία αγορά και θέλουμε την εγγύηση ότι και, τις, και τα 27 κράτη-μέλη θα μπορέσουν αποτελεσματικά να ε, ενεργούν εντός της Ευρωπαϊκής, αγορά, ε, ενός ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό ισχύει και για τη μεταφορά εμπορευμάτων και για τη διακίνηση προσώπων. Θέλουμε λοιπόν ένα core network μέχρι το 2030, απόλυτα λειτουργικό. Και η παρούσα πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ακόμη πιο φιλόδοξη, γιατί στα υπάρχοντα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών προτείνεται ένα ενδεικτικό πλαίσιο, ενώ αυτή τη φορά ζητούμε από τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δεσμεύσεις. Την υποχρέωση ότι μέχρι το 2013 συγγνώμη, θα ε, θα εφαρμόσουν αυτό το Core Network. Και αυτό προποθέτει φυσικά παιδίση μεταξύ και των 27 χωρών μελών, από όλες 27 χώρε μέλη. Έχουμε και το σχεδιασμό και ιδιαίτερε φιλοδοξίε σε θέματα σχεδιασμού. Ε, θα πρέπει να έχουμε πιο εστιασμένη και αποτελεσματική στήριξη εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και προτείνουμε να προτείνουμε μικρό αριθμό διαδρόμων Core Network, προκειμένου να συντονίσουμε τις εθνικές επενδύσεις, αλλά και τις επενδύσεις βιομηχανίας, διαχειριστών υποδομών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικές υποδομές. Πέραν του συντονιστικού ρόλου, προτείναμε και πολύ φιλόδοξο προϋπολογισμό για το χρηματοδοτικό μέσο ε, του μέσου, 31,7 δις, εκ των οποίων 10 δισεκατομμύρια είναι για τις χώρες της συνοχής. Σε ό,τι αφορά αυτά τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που αναφέρθηκαν φυσικά σήμερα το πρωί και είναι ένα από τα στοιχεία που συζητήθηκαν περισσότερο από οτιδήποτε στο μέσο συνδέοντο στην Ευρώπη και με τους ενδιαφερόμενους και με τα κράτη-μέλη, αλλά και φυσικά στην Επιτροπή σας, αλλά και γενικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά λοιπόν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπονται για χρηματοδότηση επιχορηγήσεων για το Ευρωπαϊκό Core Network και είδατε ότι στο μέσο συνδέοντα την Ευρώπη έχουμε και ένα κατάλογο με σχέδια. Οπότε τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού κατέληξαν σε περιορισμένο αριθμό σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βλέπετε από τον κατάλογο των σχεδίων ότι αυτά έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και ε, είναι ε, σιδηροδρομικά τα περισσότερα. Είναι τα πιο δύσκολα αυτά. Όχι μόνο στις χώρες συνοχής, αλλά σε όλες τις 27 χώρες. Τα διασυνοριακά τμήματα των υποδομών προσκρούν και σε τεχνικές δυσκολίες πολύ συχνά, αλλά και δεν τυχάνουν κάποιες πολιτικές προτεραιότητες. Γι' αυτό και το χρηματοδοτικό μέσο συνδέοντας στην Ευρώπη θα επικεντρωθεί κυρίως σε τέτοιου είδους σχέδια αλλά και ιδιαίτερα για αυτό το παράθυρο των 10 δισεκατομμυρίων που αφιερώνονται στις χώρες συνοχής. Και εκεί θα στηρίξουμε τις κοινέ προσπάθειες των ε, κρατών συνοχής προκειμένου να εφαρμόσουν αυτά τα πιο κρίσιμα τμήματα που είναι διασυνοριακά. Τώρα, πώς θα λειτουργήσει αυτό το μέσο. Με ανταγωνιστικές προσφορές των κρατών μελών, ένα είδος ε, πλειοδοσίας, για τα διάφορα προγράμματα εκ μέρους των κρατών μελών και φυσικά θα υπάρχει μεγάλη διαφάνεια, προβολή αυτών των σχεδίων για το ποια προγράμματα και σχέδια θα χρηματοδοτηθούν από το μέσο συνδέοντα στην Ευρώπη με το πλεονέκτημα όλα τα κράτη-μέλη, όχι μόνο οι χώρε συνοχή, αλλά όλε οι 27 χώρε-μέλη, μέχρι το 2013 που θα είναι πλήρω λειτουργικό το μέσο αυτό, να μπορέσουν να προετοιμάσουν τα σχέδιά του. Τα σχέδια αυτά ε, θα ακολουθήσουν μια διαδικασία πρόσκληση για υποβολή προσφορών, θα αξιολογηθούν με βάση την ποιότητά τους, την οριμότητα και την αποτελεσματικότητά τους, δηλαδή κατά πόσο όντως περιλαμβάνουν προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υποστήριξη μιας, ε, ενός εκτελεστικού οργανισμού και ε, επαγγελματικού εξωτερικού ελέγχου και αξιολόγηση ε, θα προκηρύξει το διαγωνισμό. Σε ό,τι αφορά αυτό το παράθυρο των 10 δισεκατομμυρίων, ο διαγωνισμό αφιερώνεται κυρίω ε, ε, και περιορίζεται στι χώρε συνοχή. Μόνο οι χώρε συνοχή δικαιούνται να καταθέσουν σχέδια για αυτά τα 10 δισεκατομμύρια. Επιπλέον, αυτά τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτήσουν κυρίως υποδομές από τον κανονισμό του Ταμείου συνοχή. Οπότε θέλουμε αυτά τα 10 δισεκατομμύρια να χρησιμοποιηθούν πλήρω για να διευκολύνουν την εθνική συγχρηματοδότηση για τέτοιου είδους σχέδια. Το βασικό σημείο της συζήτησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των διοικήσεων των χωρών της συνοχής είναι πώς η εφαρμογή και ο διαγωνισμός των σχεδίων θα εξασφαλίζουν σωστή επιλογή των σχεδίων. Δηλαδή, το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη έχει και εθνικούς φακέλους, όπως συμβαίνει με το Ταμείο της Συνοχής. Εμείς αποφασίσαμε να μην έχουμε τέτοιους εθνικούς, εθνικά κονδύλια, ε, γιατί θέλουμε να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των σχεδίων από την εμπειρία που είχαμε από τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, διαπιστώσαμε ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των σχεδίων εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα σχεδίων. Και εκτός από την ποιότητα, εξασφαλίζει και όριμα σχέδια. Και όταν επιλέγονται κάποια σχέδια TEN-T, επιλέγονται σχέδια που μπορούν άμεσα να εφαρμοστούν. Η ποιότητα και η οριμότητα των σχεδίων είναι πολύ σημαντικά στοιχεία που ασκούν και χρήσιμη πίεση στους εργολάβους των σχεδίων, στους διάφορους οργανισμούς, στους διαχειριστές των υποδομών, στα λιμάνια, σε όσους θα εκπονήσουν το σχέδιο. Και με το σύστημα αυτό μπορούμε να έχουμε ε, αναδόχους που θα υποβάλουν σωστά προγράμματα, ποιοτικά προγράμματα, που αν θέλουν να συγκεντρώσουν τους σπόρους τους, ε, θα καταφέρουν μέχρι το 2013 να υποβάλουν τα σιδηροδρομικά σχέδια και κυρίως τα διασυνοριακά για να συμπληρωθούν τα δια... ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και το Core Network. Παρόλο που δεν υπάρχουν τέτοια εθνικά, εθνική φάκελη και υπάρχει μια διαδικασία ανταγωνιστικής, ανταγωνιστικών προσφορών, αποφασίσαμε, όπως φαίνεται και στον ε, κανονισμό ε, του Ταμείου Συνοχής και στο Σύνδεδο στην Ευρώπη, όταν επιλέγουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιλέγει τα σχέδια, προσπαθεί να εξασφαλίσει μια ισορροπία ε, γεωγραφική μεταξύ των χωρών μελών. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται αυτόματα. Δεν υπάρχει αυτόματη εγγύηση, μηχανική εγγύηση για απόλυτη δικαιοσύνη στην κατανομή των σχεδίων μεταξύ των χωρών, αλλά δίνει κάποια χέγγια στα κράτη-μέλη ότι θα φροντίσουμε το Core Network και τα σχέδια που θα εμπίπτουν στο Core Network να είναι καλά κατανεμημένα μεταξύ των χωρών μελών. Και άρα το Core Network να μην εμφανιστεί μόνο σε ένα-δύο χώρες, αλλά και σε όλες τις χώρες συνοχής, αλλά και στις 27 χώρες μέλη. Να προσθέσω και να υπογραμμίσω ότι οι χώρες συνοχής έχουν ένα αποθεματικό, αυτό το το κονδύλιο των 10 δισεκατομμύριων, αλλά έχουν και πλήρη πρόσβαση και στα υπόλοιπα 21,7 δισεκατομμύρια. Στο υπόλοιπο κονδύλιο δηλαδή του χρηματοδοτικού μέσου που είναι ανοιχτό σε σχέδια από όλες τις χώρες μέλη και τι 27. Πέραν του ειδικού φακέλου, ειδικού ποσού των 10 δισεκατομμυρίων για τις χώρες συνοχής, θα προσπαθήσουμε, θα μεριμνήσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε συμπληρωματικότητα με τα υπόλοιπα μέσα, δηλαδή το Ταμείο Συνοχής ε, θα είναι διαθέσιμο για τις χώρες συνοχής και για το Core Network, για τα πιο εθνικά τμήματα του Core Network, αλλά είναι επιλέξιμο και για το συνολικό δίκτυο, ώστε να χρησιμοποιηθεί το Ταμείο Συνοχής για όλα τα, το σύστημα TEN-T και το ΕΤΠΑ να χρησιμοποιηθεί και για υποδομές και για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, αλλά και για τα επιμέρους δίκτυα των κρατών μελών που χρησιμοποιούν κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εν κατακλείδη θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η επιλογή των σχεδίων που προβλέπονται στο παράρτημα του Συνδέοντα στην Ευρώπη, η επιλογή των σχεδίων έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σε στενή συνεργασία και με τις 27 χώρες μέλη. Είχαμε πέντε γύρους διμερών συναντήσεων με τα κράτη-μέλη για να εντοπίσουμε το Core Network και τον κατάλογο σχεδίων και ιδιαίτερα για τις χώρες συνοχής και το κονδύλιο των 10 δισεκατομμυρίων. Οι συζητήσεις για τα σχέδια αυτά έγιναν από κοινού με συναδέλφους ε, της DG Radio και της DG Move προκειμένου να ενημερωθούμε για την παρούσα εφαρμογή των ε, κονδυλίων συνοχή στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, αλλά και να εξασφαλίσουμε απόλυτη συμπληρωματικότητα στην επόμενη περίοδο μεταξύ του χρηματοδοτικού μέσου συνδέοντα στην Ευρώπη και των άλλων σχεδίων που θα προταθούν από τις χώρες συνοχής για τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Και φυσικά εδώ στις συζητήσεις θα πρωτοστατήσουν οι συνάδελφοι της Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζο, αλλά φυσικά στη συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση μου, ώστε να εξασφαλίσουμε συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο μέσων. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε απορίες. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε ε, εκπροσώπους και της Γενικής Διεύθυνσης για, τη, για, για, την, για την κοινωνία της πληροφορίας και από τη Γενική Διεύθυνση ε, Ρέτζιου. Είμαστε όλοι στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε. Κύριε Διευθυντά, δίνουμε τον λόγο στον κύριο Μπερκόβιτς, πρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Έχετε λόγο. ευχαριστώ. Να πω λίγα πράγματα για τη συμπληρωματικότητα. Όπως ξέρετε, βασικό θέμα της πρότασης της Κομισιόν, του πλαισίου δηλαδή πολιετούς χρηματοδότησης, ήταν η μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των διαφόρων μέσων και βεβαίω στον τομέα των μεταφορών και ειδικά τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών αλλά και στου τομεί ε, ε, πληροφορική και τηλεπικοινωνιών και στις υποδομές ε, συνεργαζόμαστε στενά και αυτό θα είναι σημαντικό για τα κρατη στο μέλλον και οι κανονισμοί προβλέπουν δύο μηχανισμού για αυτή την συμπληρωματικότητα. Πρώτα απ' όλα είναι το κοινό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς, όπου προβλέπεται πως η Κομισιόν, αφού υιοθετηθούν όλα τα πακέτα, θα ορίσει το πόσο μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά τα θέματα στο τομέα των μεταφορών, έρευνας, εκπαίδευσης κτλ και βεβαίως ε, εδώ πέρα θα μπορέσουμε να καθορίσουμε λεπτομερέστερα τη συμπληρωματικότητα. Ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό βεβαίως είναι η εθνική πτυχή. Σε εταιρικές αυτές συμβάσεις θα δείτε πως ε, έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εδαφική ανάπτυξη και στο τμήμα αυτό έχουμε προβλέψει πως σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί για να υπάρχει συμπληρωματικότητα, συνοχή σε εθνικό επίπεδο με το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη και το τι έχει γίνει στην πολιτική συνοχή και βεβαίω θα υπάρχει μια εντατική συζήτηση μεταξύ Κομισιών και κρατών μελών για να συνεργαστούμε στον δυνατόν περισσότερο για να μεγιστοποιήσουμε την προστιμένη αξία. Και τέλο, όπω είπε και ο Νίκολα Μάρτιν, σε επιχειρησιακού όρου, ειδικά όσον αφορά μεγάλα έργα, τα οποία εξετάζει η Κομισιόν, θα συνεργαστούμε στενά με του ε, συναδέλφους μα για να διασφαλίσουμε πω όλα αυτά θα συνδυάζονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Τώρα δύο συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο, κύριο σόλγε. Ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά άκουσα τα του καλύτερου συντονισμού. Έχουμε καλά παραδείγματα από το παρελθόν, όπως παραδείγματο χάρη περιφερειακή ανάπτυξη και ανάπτυξη πέθρου. Υπέροχος συντονισμός. Βεβαίως ηρωνεύομαι, δεν γίνεται τίποτα να εκφράσω κάποια από τα στοιχεία και θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της ε, Γενικής Διεύθυνσης μου, αν κατάλαβα καλά ή όχι, γιατί είναι μια υπόθεση από ό,τι κατάλαβα. Ε, μια υπόθεση ε, κάνω και όχι μια ερώτηση. Είπατε την λέξη παράθυρο και τα λεφτά για τις χώρες συνοχής. Η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιου χρησιμοποιεί σήμερα την λέξη, τον όρο, τα λεφτά τα παίρνουμε από το Ταμείο συνοχή. Τα παίρνουμε από το Ταμείο συνοχή ή τα δίνουμε στις χώρε συνοχή. Δεύτερον, το δυσκολότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι το πλαφόν. Το λεγόμενο 2,5% του ΑΕΠ και εκεί πέρα έχουμε το Ταμείο Συνοχής. Εάν πάρετε τα λεφτά από το Ταμείο Συνοχής ή τα δώσετε στις χώρες συνοχής θα μειωθεί το πλαφόν. Και το πλαφόν θα κατέβει, αν κατάλαβα καλά, από το 2,5 στο 2,432 και τώρα έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση με τους Ούγκρους, Λετονούς και τα λοιπά και τα Οπότε το ερώτημα είναι, είναι στο πλαφόν ή όχι. Ή είναι απλά διεύρυνση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Συγγνώμη για να γίνω κατανοητός. Δεν έχω πρόβλημα με την ιδεολογία, με τη συμπληρωματικότητα. Όλα αυτά, ναι, διασυνοριακά, ωραία, κανένα πρόβλημα. Αλλά για μένα πρόκειται απλά για διεύρυνση των ευρωπαϊκών δικτύων ε, μεταφορών. Δίνουμε περισσότερα λεφτά σε αυτά και έχουμε μετά την περιχαράκωση άλλα 10 δισεκατομμύρια για τις χώρες ε, της συνοχής. Ε, να το πούμε με το όνομά του και αν συμφωνούν τα κράτη-μέλη να πέσει το πλαφόν, εντάξει. Άλλο θέμα. Ολόκληρη η πολιτική συνοχή βασίζεται στη μεθοδολογία που ανέφερε ο κύριος Μποστινάρου περί κοινή διαχείρισης. Εάν τα λεφτά τα πάρετε από το κομμάτι της συνοχής ή τα δώσετε στις χώρες συνοχής, το ερώτημα είναι θα έχουμε κοινή διαχείριση με ό,τι συνέπειες έχει αυτό για τον κανονισμό ή θα είναι κάτι κεντρικό από τις Βρυξέλλες στο, σε μια ε, υπηρεσία, αν δεν ξοδευτούν τα λεφτά, Ποιο θα είναι ο υπεύθυνο. Ε, η υπηρεσία ή τα κράτη-μέλη. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί είτε ε, μιλάμε για κοινή διαχείριση ή προσθέτουμε κάτι το νέο. Έχω, δεν έχω πρόβλημα. Ας δώσουν περισσότερα λεφτά στα ευρωπαϊκά δίκτυα, στα συνοριακά. Η άλλη ιδέα δικτυα σταδια συνοριακα η αλλη ιδεα ειναι να τα αφήσουμε στο Ταμείο Συνοχής στον εθνικό φάκελο, γιατί έχετε δίκιο. Δεν υπάρχουν εθνικοί φάκελοι στην υπηρεσία, αλλά υπάρχουν εθνικοί φάκελοι στην πολιτική συνοχή. Ε, δεν μπορούμε να τα ανακατεύουμε όλα. In the, national envelopes, we can earmark... Ε, αν τα αφήσουμε λοιπόν στο εθνικό φάκελο, μπορούμε να τα δεσμεύσουμε και θα είναι αναγκασμένα να κάνουν τα κράτη-μέλη το έργο που έχει αποδεχτεί η υπηρεσία θα είναι το ίδιο, αλλά βεβαίω η ευθύνη θα ανοίξει τα κράτη-μέλη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, δεν έχω τίποτα κατά του μέσου αυτού. Τίποτα κανένα πρόβλημα με την ιδεολογία, διασυνοριακές συνδέσει και να ονειρευόμαστε περί συμπληρωματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Είναι, είναι όνειρο εδώ μέσα, αλλά όσον αφορά τη μεθοδολογία και τις πολιτικές συνέπειες, τα πράγματα θα είναι δύσκολα γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά εάν τα λεφτά τα πάρουμε παραδείγματο χάρη από τον πολωνικό φάκελο του Ταμείου Συνοχής και τα πάρουν από, τους Ρουμα, από το ρουμανικό φάκελο και η Πολωνία θα κερδίσει θα πάρει τα πολωνικά λεφτά τι θα πούν οι Ρουμάνοι θα πούν μας πήρατε τα λεφτά μας μπορεί να κάνω λάθος αλλά ξεκαθαρίστε το γιατί εμείς είμαστε πολιτικοί και πρέπει να απαντήσουμε σε αυτά που μας λέει ο κόσμος. Τι κάνουμε, υπερασπίζουμε τους εθνικούς φάκελους ή τους μειώνουμε. Ε, έχει σημασία αυτό, καταλαβαίνετε, από πολιτική σκοπιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας υπενθυμίσω πως πρέπει να τελειώσουμε σε 11.30 για να έχουμε και λίγο χρόνο στον εκπρόσωπο. Παρακαλώ λοιπόν ερωτήσεις. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Α, ερωτήσει. Σε αντίθεση με τον συνάδελφο, τον κύριο Όλμπριχτ, εγώ έχω σοβαρέ αμφιβολίε για την αποτελεσματικότητα του μέσου αυτού που υποτίθεται πως θα έχει και ε, δικές της αρχές γιατί ξέρετε πως ε, το καλύτερο είναι εχθρός του καλού και μιλάμε ότι είχε προβλεφθεί να χρηματοδοθεί αμέσως 40 δισεκατομμύρια και άλλα 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής. Αυτό είναι μόνο μια πτυχή. Θεωρώ πως είναι αποτέλεσμα της συζήτησης που είχαμε το εάν υπάρχει πολιτική συνοχή ως περιφερειακή πολιτική ή τομεακή πολιτική. Και για να καθησυχάσω δε, τους τομεακούς εδώ μέσα, είχαμε πει πώς θα επικεντρωθούμε στην ενέργεια, συγκοινωνίες και τηλεπικοινωνίες για να δώσουμε και λίγα λεφτά στρατηγική του 2020 μόνο που από τη συζήτηση στην Επιτροπή ε, Συγκοινωνιών όπου είμαι αναπληρωματικό μέλος και είχαμε συζήτηση για την εφαρμογή των έργων των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και των υποδομών δεν έχω πιστεί εγώ πως θα καταφέρουμε αυτό το οποίο θέλουμε εδώ πέρα. Τα προβλήματα διασύνδεσης των μεγάλων σιδηροδρομικών δικτύων στην Ευρώπη δεν είναι κατά βάση προβλήματα χρημάτων, αλλά προβλήματα προκύπτουν από το ότι ο καθένας ε, στις 27 χώρες φτιάχνει το δικό του τρενάκι και δεν ε, κάνουν ε, τυποποίηση. Τι να σας πω τώρα, από τη σήμανση, το τροχαίο υλικό, τα διαφορετικά βολτ στο ηλεκτρικό δίκτυο των γραμμών, και άμα μιλάμε δηλαδή για διασυνεριακή συνεργασία και τα λοιπά για να ξεπεράσουμε τις ε, στενοπούς, τότε νομίζω πως ε, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει ανταγωνισμός διαφορετικών σιδηροδρομικών ε, εταιριών και τα λοιπά, Το ίδιο και με την ενέργεια. Εδώ πέρα πρέπει να δράσουν τα κράτη-μέλη. και βεβαίως ε, θα πρέπει να δούμε και την ε, κοινωνική πτυχή, όχι μόνο το τι θέλει ένα κράτος μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ πέρα βεβαίως έχουμε το πρόβλημα πως ε, διασυνοριακά γίνονται λίγα πράγματα όσο δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια εσωτερική αγορά ενέργειας. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε προβλήματα μεθοδολογίας παρά οικονομικά και κατόπιν όσον αφορά την ευρυζωνικότητα ή ευρυζωνικότητα. Είναι θέμα των τηλεπικοινωνιακών εταιριών σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Τι θα κάνουμε, θα τους δώσουμε τώρα οικονομική στήριξη για να συνδέσουν περιοχές με ευρυζωνική σύνδεση εκεί όπου δεν τους συμφέρει. Και τέλος, που είπε για τη διαφάνεια και την διοίκηση, τη διαχείριση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη παρά το ότι σε πολλές περιπτώσεις τα κράτη-μέλη μόνο έμεσα είναι υπεύθυνα για αυτές τις υποθέσεις. Επίσης ε, και οι περιφέρειες ε, όταν αναζητούν μόνες τους λύσεις ε, έχουν την δυνατότητα βεβαίως να αναζητήσουν κάποια μέσα για να κάνουν μικρότερα έργα. Βεβαίως αυτό πάλι ε, θα είναι σε αντίφαση με τα μεγάλα διασυνοριακά έργα διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Οπότε εδώ πέρα προκύπτουν πολλά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με την πρόταση αυτή κανονισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποστινάρου έχει το λόγο. Chairman, thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να προσθέσω καινούριε προκλήσεις μετά από τον αγαπητό συνάδελφο κύριε Όλμπραϊτ. Ανέφερε αρκετές. Ε, ως έννοια, μάλλον επί της αρχής δεν έχω καμία αντίρρηση. Μια διασυτοριακή ε, υποδομή που θα μας επιτρέψει να έχουμε την Ευρώπη ως μια ενιαία ονότητα όπως συσχύει στις Ηνωμένε Πολιτείε ή στην Κίνα, να έχουμε αυτά τα μεγάλα έργα υποδομής. Αλλά ο διάβολος βρίσκεται στη λεπτομέρεια. Και η απάντησή σας δεν μας δίνει ίχνος απτής πληροφορίας για τις λεπτομέρειες. Εδώ, τίποτε για το πώς θα γίνει. Γιατί πώς θα γίνει σημαίνει χρήματα. Πόσα χρήματα θα χάσει το ένα κράτος μέλος για να τα κερδίσει κάποιο άλλο κράτος μέλος στην περίπτωση που ε, ένα κράτος μέλος ε, ε, για παράδειγμα, η Ρουμανία χάσει έναντι της Πολωνίας στο σενάριο που ανέφερε ο κύριος Ολβράχτ. Έχουμε κάποιο σενάριο για τους νικητές και τους ιτημένους και όχι μόνο για τις χώρες αλλά και για τις επιχειρήσεις. Γιατί όταν χάνεις εκατομμύρια η χώρα που θα χάσει τα εκατομμύρια θα χάσει και τις συμβάσεις και τις υπεργολαβίες και αυτό θα δημιουργήσει ε, απογοήτευση. Είμαστε πολιτικοί μας ενδιαφέρουν οι ψηφοφορίες, οι εκλογές, οι χώρες που χρειάζονται περισσότερα από άποψη υποδομής, μερικές φορές έχουν πολύ μικρή, χαμηλή, φτωχή διοικητική ικανότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ε, προγράμματα μεγάλης κλίμακας. Ε, θα πρέπει λοιπόν τώρα να φανταστούμε ποιοι ενδεχομένως θα χάσουν. Έχουμε κάποιο φάρμακο για αυτό το πρόβλημα. Γιατί όταν γυρίσουμε πίσω θα πρέπει να εξηγήσουμε όχι μόνο στη Ρουμανία αλλά και στους συναδέλφους. Ε, πρέπει ε, τι θα γίνει με τις χώρες της Παραδονάβιες, τις Βαλτικές. Ε, όλοι συζητούμε μεταξύ μας ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις για τις πολιτική συνοχής. Και δεν είναι και δική μου ανησυχία μόνο, είναι και δική τους ανησυχία. Πρέπει να πείσουμε τις κυβερνήσεις να το κάνουν, να το δεχθούν. Αλλά για να το δεχθούν χρειάζεται να έχουμε μία δίκαιη ισορροπία. Και τέλος, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μας, ζητάτε τώρα να σας δώσουμε μία επιταγή εν λευκό. Για να δούμε το 2014 ποια έργα θα επιλεγούν μετά από τη του χρηματοδοτικού, μετά από την ψήφιση του πολιετούς χρηματοδοτικού πλαισίου. Ζητάτε τώρα από μας πλήρης εγγύησης όταν εμείς δεν έχουμε καμία εγγύηση για τη δικαιοσύνη του σχεδίου, για τον αντίκτυπο του χρηματοδοτικού μέσου συνδέοντας την Ευρώπη σε κάθε κράτος μέλος. Γιατί η πολιτική συνοχή εν τέλει συνίσταται στην αποκατάσταση ανισοτήτων, ε, όχι στην δημιουργία νέων ανισοτήτων. Και η απάντησή σας δεν είναι ικανοποιητική για να το θέσω έτσι. Εμείς θέλουμε να ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη. Ποια προγράμματα συζητάτε αυτή τη στιγμή με τα κράτη-μέλη. Τα πιο σημαντικά διακρατικά προγράμματα υποδομής τα οποία συζητούμε και τα οποία θέλουμε να τονώσουμε με το χρηματοδοτικό μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Χωρίς πληροφορίες, χωρίς ενημέρωση, μα εικάζουμε, οικοτολογούμε. Κοιτάξτε, είμαστε πολιτικοί και πριν να ψηφίσουμε χρειαζόμαστε κι εμείς εγγυήσει. Όχι, δεν σας δίνουμε επιταγές εν λευκό. Όχι τέτοιες σχέσεις μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κωστινάρου. Ε, ποιος αντιπρόσωπος της ε, Επιτροπής θα απαντήσει. Ίσως εγώ θα έπρεπε να αρχίσω, αν δεν σας πειράζει. Και ο Πίτερ θα μιλήσει για τα πλαφόν. Νομίζω ότι είναι πιο αρμόδιος από μένα. Γι' αυτό. Οι τιμένοι και νικητές χαμένοι και νικητέ, Νομίζω ότι ο στόχο ο ίδιο του χρηματοδοτικού μέσου είναι να στηρίξει την ένταξη των χωρών στην ενιαία αγορά. Περί αυτού πρόκειται. Χωρίς να επικεντρωθούμε, χωρίς ε, οι προσπάθειε των κρατών μελών να επικεντρωθούν και σε και όλες εκείνες οι χώρες που έχουν διακρατικά συμβάσεις και έργα αυτή τη στιγμή, δεν συμβαίνει σήμερα ούτε στις χώρες συνοχής, ούτε σε όλα τα 27 κράτη-μέλη. Και εδώ ε, μέρος του σχολιασμού σας ε, είναι έγκυρος. Πράγματι το ρυθμιστικό πλαίσιο, τα διακρατικά έργα δημιουργούν κάποια κυβερνητικά εμπόδια, αλλά το πλαίσιο προγραμματισμού πρόκειται να τα επιλύσει αυτά. Έχουμε προτείνει κανονισμούς όχι μόνο για τα κράτη-μέλη, για τον διαχειριστή της υποδομής, για τις σιδηρόδρομους κτλ. Λοιπόν, οι κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετωπίζουν το θέμα των κυβερνητικών εμποδίων, τα προγράμματα θα οριμάσουν, αλλά χρειαζόμαστε περαιτέρω όθηση και το χρηματοδοτικό μέσο συνδέοντας την Ευρώπη μας παρέχει αυτή την όθηση. Πιστεύω ακράδαντα ότι εξασφαλίζοντας πρόσβαση στην ε, εσωτερική αγορά για τις χώρες συνοχής, συμβάλλουμε, χτίζουμε τη συνοχή. Συμβάλλουμε διασφαλίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη θα υπάρξει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι το μόνο και πιο αποτελεσματικό εργαλείο που έχουμε, αλλά είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη. Και επανέρχομαι στο πραγματικό ερώτημα που το, και ε, για το θέμα χαμένων και νικητών μεταξύ των κρατών μελών και πώς λειτουργεί. Ε, δεν σας είπα αρκετά πράγματα. Ίσως τώρα μπορώ να γίνω λίγο πιο ακριβής. 29 και 30 Νοεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, διοργανώνουμε ένα συνέδριο ε, για την ε, προσέγγιση και θα μιλήσουμε ακριβώς για τις λεπτομέρειες του πώς το χρηματοδοτικό μέσο συνδέοντας σε την Ευρώπη θα κινηθεί σε αυτό το παράθυρο των 10 δισεκατομμαρίων. Ε, είσαστε ευπρόσδεκτοι. Ε, μπορούμε να έχουμε και διμερείς συναντήσεις ή αν θέλετε και ένα πιο αναλυτικό σεμινάριο να οργανώσουμε για να σας δείξουμε πώς η Εκτελεστική Επιτροπή των Διευρωπαϊκών Δικτύων επιλέγει και διαχειρίζεται τα έργα και πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει μέγιστο αντίκτυπο για τα προγράμματα και επίσης για το ότι τα προγράμματα είναι έτοιμα στην ώρα τους. Για να απαντήσω την ερώτησή σας για τους χαμένους και τους νικητές. Καταρχήν πολιτικά δεν θα υπάρξουν χαμένοι. Η όλη ιδέα είναι να φέρουμε κοντά τα κράτη-μέλη. Ο τρόπος που θα λειτουργήσουμε είναι ο εξής. Το 2011, 2012 και 2013 τα 10 διευρωπαϊκά προγράμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα χρηματοδοτικά μέσα της ε, πολιτικής συνοχής θα διατεθούν για την προετοιμασία των έργων. Ναι, έχετε δίκιο λοιπόν. Υπάρχει, υπάρχει διαφορετική διοικητική ικανότητα μεταξύ των κρατών μελών για το χειρισμό. Ε, θα καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια με τα κράτη σε δυσκολίες να ετοιμαστούν και να καταρτιστούν τα προγράμματα που βλέπετε στο παράρτημα του χρηματοδοτικού μέσου συνδέοντα στην Ευρώπη. Υπάρχουν και χρηματοδοτικά μέσα στα οποία συμβάλλει και το Κοινοβούλιο μέσω τη διαδικασία συναπόφαση. Έχουμε δυόμιση χρόνια για να προετοιμάσουμε σε όλες τις χώρες συνοχής δεν θα καθίσουμε να περιμένουμε ποια είναι καλά και ποια δεν είναι καλά. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει το δίκτυο. Όχι να δούμε ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό κτλ. Θα συνεργαστούμε με όλους λοιπόν και θα καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια εκεί που υπάρχουν ασθενείς διαχειριστές της υποδομής των υποδομών. Επίσης, τα κράτη-μέλη ε, θα υποβάλουν προτάσεις το 2014, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια προγραμματισμού θα έχουμε ίσως δύο ή τρεις προκηρύξεις ε, για την υποβολή προτάσεων. Και αν δεν είναι όλα έτοιμα μέχρι το 2014, θα υπάρξει και δεύτερη και τρίτη παράταση. Πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Θα υπάρξει εξωτερική αξιολόγηση, ε, εκτελεστικός φορέας, ο οποίος θα εξετάσει την ποιότητα των έργων, των σχεδίων. Και δεν είναι πολιτική έρευνας όπου θα κατατάξουμε ε, τα προγράμματα ανάλογα με το ποιο είναι καλύτερο. Όχι, δεν το κάνουμε αυτό. Η εξωτερική αξιολόγηση περιλαμβάνει κάποια ελάχιστα κατόφλια ποιότητας, ορίμανσης και σημασίας. Τρία από πέντε. Αυτό επιτρέπει στο φορέα να μας πει ποια έργα δεν είναι έτοιμα για χρηματοδότηση και όταν δεν είναι, δεν έτοιμα κάποια έργα για χρηματοδότηση, υπάρχει δεύτερος και τρίτος κύκλος προκηρύξεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΜΟΥΒ, αλλά και η Ρέτζιο για το παράθυρο των 10 δισεκατομμυρίων θα εξετάσουν τα καλά προγράμματα, όχι μόνο τα εξαιρετικά. Μέσα από τη φάση προπαρασκευής και μέσα από αυτό το μηχανισμό, ξέρω από την εμπειρία μου ότι θα έχουμε έργα σε όλα τα κράτη-μέλη. Και στη συνέχεια με βάση τις διατάξεις του Ταμείου Συνοχής ε, και της ε, δαφικής συνεργασίας. Τέλος πάντων δεν ξέρω ποια είναι η ακριβής γλώσσα. Θα σας τα διαβάσω. Θα δώσουμε την μεγαλύτερη δυνατή προτεραιότητα σε έργα που έχουν εθνική ε, διάθεση πόρων. Εμείς θέλουμε να βγούμε όμως από αυτή την εθνική λογική και να εστιάσουμε στην συνδικτύωση και ιδιαίτερα στα διακρατικά διασυνοριακά έργα. Και όλοι το είπατε σαφώς και η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση, θα συνεργαστούμε και αυτό είναι και το θέμα της όλη μας πολιτικής. Θέλουμε σε όλες τις χώρες συνοχής να υπάρξει. Δεν θέλουμε τα 10 δισεκατομμύρια να πάνε σε δύο μόνο χώρες συνοχής. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να προάγουμε την ε, κατασκευή αυτού του μηχανισμού, σε, το, το, των έργων υποδομής σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι εθνικό ε, κονδύλιο. Έχετε δίκιο. Ωστόσο, με όλη τη διαδικασία, με την πολιτική δέσμευση με το, με, που αντανακλάται στον κανονισμό, υπάρχει πολιτική εγγύηση ότι τα έργα θα χρηματοδοτηθούν σε όλες τις χώρες. Για μένα λοιπόν δεν υπάρχει νικητής και δεν υπάρχει χαμένος. Πώς θα λειτουργήσει τώρα στη συνέχεια όσο αφορά τη διαχείριση των ε, έργων. Πολύ σημαντικό και αυτό το ζήτημα. Και θα υπάρξει, θα συνεχιστεί το σημερινό σύστημα διαχείρισης των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Υπάρχει η επιλογή των έργων. Αυτό δεν γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνεται και με τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα από κοινού. Και αφού επιλεγούν τα έργα, ο, ο, φορέας και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς μαζί με τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν επί της χρηματοδότησης με βάση αυτά που σας είπαμε στην πρόταση και με βάση όσων έχουν αποφασιστεί και σχεδιαστεί κατά τη διαδικασία προετοιμασίας. Μετά υπάρχει η πρώτη καταβολή, ε, η πρώτη αποδέσμευση κονδυλίων. Αυτό συμβαίνει προοδευτικά καθώς προχωράει η υλοποίηση του έργου όλοι γνωρίζετε αυτόν τον τρόπο διαχείρισης και η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο το κάνει λίγο διαφορετικά, αλλά ε, εάν, εν πάση περιπτώσει, το έργο δεν προχωράει, τότε μειώνεται η χρηματοδότηση. Δύσκολη είναι αυτή η αρχή. Το κάναμε για πρώτη φορά το 2010 Κατά την αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου, τα κράτη-μέλη δεν ένιωσαν και τόσο καλά. Και τα 27, έτσι, γιατί υπάρχουν τέτοια ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών παντού. Αλλά με αυτή την ε, ε, αρχή, ή, τα παίρνεις ή τα χάνεις, δημιουργείται πολιτική ε, πίεση. Και δημιουργεί αποτελέσματα στην υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Έτσι γίνεται η διαχείριση από τον φορέα για που αποφασίζει για τα μέσα χρηματοδότησης. Αν δεν χρησιμοποιηθούν οι πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος, δεν χάνονται, επανέρχονται, επιστρέφουν στο πρόγραμμα και επαναδιοχετεύονται σε προκηρύξεις. Και πάλι λοιπόν κάνοντας την επιλογή ε, δουλεύουμε πάνω στην εθνική κατανομή των πόρων. Έχουμε υψηλό βαθμό λοιπόν προβλεψιμότητας με βάση τον κατάλογο των έργων, τη δέσμευση της Επιτροπής να δουλέψει πάνω στα εθνικά κονδύλια. Από την ίδια στιγμή ο ανταγωνισμός μεταξύ των έργων εξασφαλίζει την ορίμανση και την ε, ετοιμασία τους στην ώρα τους. Βεβαίως η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι λαμβάνονται οι αποφάσεις χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια η υλοποίηση στο πεδίο, ε, δημόσιες συμβάσεις, ανάθεση κτλ. Αυτό ανήκει στα κράτη-μέλη όπως γινόταν μέχρι στιγμή. Στις χώρες συνοχής συχνά είναι η ίδια διοίκηση η οποία αναφέρεται προς την οφορέα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα κάθε δύο χρόνια και επιβεβαιώνει κατά πόσο υπάρχει ανάγκη περαιτέρω χρηματοδότησης. Είναι λοιπόν ένα πολύ συγκεντρωτικό σύστημα όσο αφορά την επιλογή, τη χρηματοδότηση, αλλά είναι σχετικά παρόμοιο ε, με το σύστημα συνοχής όσο αφορά την υλοποίηση. Έτσι λοιπόν στην Επιτροπή αναμένουμε ότι τα κράτη-μέλη ήδη έχουν τους θεσμούς, τα όργανα και την ικανότητα για να λειτουργήσουν και να τρέξουν το πρόγραμμα. Λοιπόν, το παράθυρο των 10 δισεκατομμυρίων. Το χρηματοδοτικό μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Ε, Γενική Διεύθυνση Ενέργεια, MOVE, Regio θα, και οι τρεις αυτές γενικές διευθύνσεις θα υλοποιήσουν το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Δεν έχουμε αποφασίσει πώς ακόμα, αλλά σε αυτό, πάνω σε αυτό εργαζόμαστε. Βεβαίως το ερώτημα είναι από πού θα προέλθουν τα δισεκατομμύρια. Προφανώς και έρχονται από το Ταμείο Συνοχής. Ναι. Ο συνάδελφος θα απαντήσει σε ένα λεπτό. Θα μεταφερθούν λοιπόν σε ετήσια βάση. Ο κανονισμός είναι σαφής. Ετησίω θα μεταφέρονται τα κονδύλια αυτά. Η επιλογή για αυτή τη μεταφορά υπαγορεύθηκε και από την απόφαση της Επιτροπής να τα κρατήσει για τις χώρες συνοχής. Αυτή είναι η λογική της μεταφοράς. Τα χρήματα δεν τα παίρνουμε από τις χώρες συνοχής. Δεν ισχύει. Μεταφέρονται σε μια ελαφρώς διαφορετική διαχείριση. Γιατί τα έργα αυτά είναι διαφορετικά προγράμματα και αυτό δικαιολογεί τη διαφορετική διαδικασία διαχείρισης, αλλά θα υλοποιηθούν προς όφελος και με τις χώρες εργαζόμενοι πάνω στα εθνικά κονδύλια, τα εθνικά χαρτοφυλάκια, προς την ολοκλήρωση της αγοράς. Νομίζω λοιπόν ότι εν τέλει εποφελείται η συνοχή. Και τώρα ο συνάδελφος. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Ο κύριος Μπέργκοβιτς θέλει να κάνει κάποια σχόλια. Παρακαλώ όμως, επειδή έχουμε ξεπεράσει τα χρονικά όρια, να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντομος γίνεται. Θα είμαι ε, λακωνικότατος. Σε ό,τι αφορά τους σαφείς μηχανισμούς δημοσιονομικής τεχνικής ε, και το θέμα της κατάρτισης του προϋπολογισμού για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, σας παραπέμπω στους συναδέλφους Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμών. Αλλά εγώ θα μιλήσω για το μηχανισμό που περιλαμβάνει ο κανονισμός μας. Οι εθνικοί φάκελοι, τα εθνικά ποσά για τα, από το Ταμείο Συνοχής θα συστηθούν και θα υπολογιστούν με βάση το MFM θα γίνουν γνωστά τα ποσά κατά το τέλος της συζήτησης και τα ποσά αυτά θα υπόκειται στο πλαφόν ως τμήμα του συνόλου. Το ποσό των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που προβλέπεται για το μέσο συνδέοντα στην Ευρώπη για τις χώρες συνοχής θα αφαιρεθούν. Θα είναι προοράτα από τους εθνικούς φακέλους. Δηλαδή τα 10 δισεκατομμύρια θα οδηγήσουν σε μείωση 15% αλλά η ίδια μείωση θα ισχύσει για όλα τα κράτη-μέλη. Του Ταμείου Συνοχής, του κονδυλίου της, το κονδυλίο της Συνοχής. Κατόπιν θα, φυσικά το ποσό θα υπολογιστεί για το σύνολο της περίοδου, για ολόκληρη την περίοδο και θα μεταβιβαστεί στον προϋπολογισμό του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη για, στη δημοσιονομική γραμμή που προβλέπει εφαρμογή των διευρωπαϊκών δικτύων ε, μεταφορών. Κατόπιν θα υπολογίσετε με βάση τις αιτήσει πιστώσεις και φυσικά θα, θα είναι ιδιαίτερα αφιερωμένα στις χώρες συνοχής και θα δίνεται προτεραιότητα στα εθνικά προγράμματα και η μεταχείριση, η αντιμετώπιση είναι ίδια. Το πλαφόν, το κάπινγκ δεν αλλάζει. Αυτό δεν ε, αλλάζει, ισχύει όπως ίσχυε και προηγουμένως. Καλώς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση του μέσου αυτού και τις απαντήσεις. Και πέραμε τώρα στο επόμενο σημείο, το σημείο 14, που προβλέπει παρουσίαση της εξωτερικής μελέτης με θέμα τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα των διαρθρωτικών ταμείων και των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που απευθύνονται στι μικρομεσαίε επιχειρήσει των διαφόρων περιφερειών. Η παρουσίαση θα γίνει από την κυρία Χέρτα Τέντλινγκ Σενχόφερ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με ακούτε καλά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας ανέθεσε μία μελέτη Δεν είμαι σίγουρη ότι η φωνή μου είναι αρκετά στεντόρια για να υπερισχύσει τι πασαρίε. Λοιπόν, μα ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη διεξαγωγή μια μελέτη για τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα των διαρθρωτικών ταμείων και των ευρωπαϊκών πολιτικών που απευθύνονται προ μικρομεσαίε επιχειρήσει στι διάφορε περιφέρειε. Καταρχήν δεν πρόκειται για αξιολόγηση το ζητούμενο της ε, μελέτης είναι τι μπορούμε να πούμε για τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τα διάφορα έγγραφα για τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών και των διαρθρωτικών ε, κονδυλίων. Έχω μια τομεακή πολιτική και έχουμε κάποια στοιχεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποια είναι η φύση και τι παράγοντες επηρεάζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολλές φορές προβάλλονται ως η λύση για, τις, για την απασχόληση. Περιέχουν το μεγαλύτερο δυναμικό δημιουργία θέσεων εργασία. Τι γνωρίζουμε γι' αυτό. Επίση, πώ τα κοινοτικά όργανα ε, στηρίζουν και ευνοούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το βασικό θέμα της μελέτης είναι πώς συμβάλλει η πολιτική συνοχή στη στήριξη των μεσαίων επιχειρήσεων και τι συμπεράσματα μπορούμε να αντλήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια σύντομη ε, εξέταση αυτών των πέντε σελίδων. Καταρχήν, ως προς τη φύση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπάρχει κάτι απλό και αυτονόητο σχεδόν, αλλά που δεν αναφέρεται συχνά. Οι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μια γενίκευση. Ε, λέει ο κινητικός ορισμός πρέπει να έχει λιγότερο από 250 εργαζόμενους, λιγότερο από 50 εκατομμύρια ε, ε, γύρω εργασιών και λιγότερο από 43 εκατομμύρια στο ισοζύγιο ε, στοιχεία του ενεργητικού. Οπότε έχουμε μπορεί τις κομμωτές, να, έχουμε, να είναι οι επιτερίες αυτές από κομμωτές, κομμωτικές, ή ε, κατασκευής παπουτσιών με μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 100 εργαζόμενου. Είναι ευρύτατο δηλαδή ο κοινοτικό ορισμό για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και δεν αντανακλά πιστά αυτό το ευρύ φάσμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το θέμα είναι πώ θα περιγράψουμε καλύτερα τι εστί μικρομεσαία επιχείρηση. Το πρώτο στοιχείο είναι σαφέ. Υπάρχει διαφορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάλογα με το βιομηχανικό κλάδο στον οποίο ανήκουν, ανάλογα με την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Μπορεί να έχουν επιστημονική βάση να δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες, να ασχολούνται με τη γεωργία, να ασχολούνται με την πληροφορική και τις επικοινωνίες. Ευρύ είναι το φάσμα των δραστηριοτήτων. Άλλη διαφοροποίηση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να είναι μια νεοπαγής επιχείρηση ή μπορεί να είναι μια όριμη επιχείρηση. Οπότε είναι και διαφορετικές οι ανάγκες της επιχείρησης ανάλογα με το σε τι φάση ε, λειτουργίας βρίσκεται μια πιο όρημη επιχείρηση, οι ανάγκες ε, των παρεμβάσεων είναι πολύ μεγαλύτερες. Ενώ στην... όταν η επιχείρηση βρίσκεται στα σπάργανα, αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι χρηματοδότηση, κονδύλια, ιδέες, τεχνολογία. Αργότερα θα χρειαστούν οργανωτικές δεξιότητες και διαχειριστικές ικανότητες για να γιγαντωθεί αυτή η επιχείρηση και να ανταπεξέλθει στο σκοπό της. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που είναι σκόπιμο να το λάβουμε υπόψη. Πολύ συχνά βλέπουμε στη βιβλιογραφία ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, δεν προσπαθούν καν να, να μεγαλώσουν για να αποφύγουν τις περισσότερους κινδύνους. Ε, επίτηδες εσκεμμένα μένουν σε μικρές διαστάσεις και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ασχολούνται με καινοτομία η έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Από τις 100 μικρομεσαίες, μόνο 30 έχουν κάποια σχέση ή εφαρμόζουν κάποια στρατηγική που σχετίζεται με την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη. Και μόνο 3% έχουν υψηλέ επιδόσει στο τομέα αυτό. Η συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν εμπίπτει στην ε, κατηγορία της στήριξης για λόγους καινοτομίας. Σε ό,τι αφορά τον κύκλο της ζωής μιας επιχείρησης, βλέπουμε ότι στην αρχή αυτό που βοηθάει μια επιχείρηση είναι οι ιδέες. Αλλά όταν βλέπουμε ποιοι είναι οι πιο κρίσιμοι παράγοντες, βλέπουμε ότι στην πορεία της επιχείρησης χρειάζονται ηγετικές ικανότητες, διαχειριστικές ικανότητες, αυτές θα καθορίσουν την οργάνωση της επιχείρησης και την πρόοδο της επιχείρησης. Δεν είναι σαφές λοιπόν το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις. Όταν προσπαθεί κάποιος να χρηματοδοτήσει ή να βοηθήσει μια μικρομεσαία επιχείρηση, τι λαμβάνει υπόψη. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Ε, υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες, ε, κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον, ε, περιβάλλον, οικονομικό περιβάλλον της αγοράς, επιτόκια, εμπόριο, ε, ακόμη και το πολιτικό, θεσμικό, κανονιστικό πλαίσιο, όλα αυτά επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, είναι εξωτερική παράγοντες, αλλά υπάρχουν και εσωτερικοί παράγοντες. Για παράδειγμα, δεξιότητες διαχειριστικές και το κεφάλαιο φυσικά. Εκεί χρειάζονται πολλές φορές στοχευμένες παρεμβάσεις και φυσικά ανθρώπινη πόρη, ανθρώπινο δυναμικό και η θέση της μικρομεσαίας επιχείρησης στην αγορά. Δεν θα ήθελα να περιπλέξω εδώ την παρουσίαση, απλώς θα ήθελα να σας δείξω ότι δεν είναι εύκολο να λέμε έχουμε ένα μηχανισμό ή ένα μέσο που στοχεύει, απευθύνεται προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απευθύνεται στην καινοτομία. Και εδώ έχουμε πολλές κατηγορίες και εδώ έχουμε και εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες που επίσης διαφέρουν ε, ανάλογα με το σε ποια φάση της ανάπτυξης της βρίσκεται μια επιχείρηση. Σας παραπέμπω στην έκθεση που είναι πολύ πιο διεξοδική ως προς τα στοιχεία αυτά. Επίσης, όταν εξετάζουμε τα, διαφορα, τα διάφορα μέσα στήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπιστώνουμε ότι και εδώ έχουμε πολλά είδη παρεμβάσεων ε, στην ανάπτυξη και μεγέθυνση μιας ε, μικρομεσαίας επιχείρησης. Καταρχήν, ρυθμιστική ε, υποστήριξη. Τι μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το Small Business Act που προβλέπει κάποιες αρχές για κοινοτικές και εθνικές πολιτικές δίνοντας έμφαση στη λήψη υπόψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βέβαια, αυτή η πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις δεν αντικατοπτρίζει ούτε την περιπλοκότητα, ούτε την ποικιλομορφία, αλλά ούτε και τις ε, διαφορετικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά μπορούμε να ε, κατατάξουμε αυτές, αυτά τα μέσα στήριξης σε κανονιστικά μέτρα, ρυθμιστικά, που δίνουν ε, κάποιε κατευθυντήριες γραμμές, σε χρηματοοικονομικά, ε, χορήγηση επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, δανείων, Μερικές φορέ αφορούν την καινοτομία αυτά τα μέσα, άλλες φορές έχουν σχέση με το περιβάλλον, τον πολιτισμό ή άλλου τομεί. Έχουμε παροχή συμβουλών, συμβουλευτικά μέσα δηλαδή και στήριξη και επίσης ε, τη δικτύωση και συμμετοχή. Όλα αυτά τα μέσα είναι σχετικώς ε, ανεξάρτητα από την πολιτική συνοχή. Ελάχιστη είναι οι δεσμοί και οι στόχοι με την πολιτική συνοχή. Όταν διαρωτόμαστε λοιπόν τι κάνει η πολιτική συνοχή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διαπιστώνουμε ότι οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές μας δίνουν διάφορες πληροφορίες. Λέμε, επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας, προσελκύοντας ε, ε, στο επιχειρηματικό περιβάλλον τον κόσμο, προωθούν την καινοτομία, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία της πληροφορίας, στηρίζουν τις επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι Υπάρχουν σαφείς στόχοι για το με ποιο τρόπο η πολιτική συνοχή απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά γενικά. Όταν όμως γινόμαστε πιο σχολαστικοί και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε πώς απευθύνεται η πολιτική συνοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ποια είναι τα κονδύλια που προβλέπει για το σκοπό αυτό, τότε βλέπουμε ότι περνάμε στο επίπεδο της επέμβασης. Βλέπουμε τι κάνει το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τι κάνει το Ταμείο το κοινωνικό ταμείο. Βλέπουμε τους κώδικες παρέμβασης και εκεί διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τρία είδη παρέμβασης. Μέσα που στοχεύουν στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως το RTT, δηλαδή επενδύσεις που σχετίζονται με την έρευνα. Υπάρχει η στήριξη γνήσια υπηρεσία ε, της επιχειρήσης και επίσης αναδιάρθρωση και προσαρμοστικότητα των εργαζομένων έχουμε το παράρτημα 4 του Γενικού Κανονισμού, στο οποίο κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα προβλέπει συγκεκριμένα κονδύλια για αυτούς τους στόχους. Άμεση και έμεσης υποστήριξη. Αυτή είναι τώρα η προσέγγιση. Αλλά ποιο είναι το δίδαγμα που μπορούμε να αντιλήσουμε. Δηλαδή, με ποιο τρόπο τα κοινοτικά μέσα και κυρίως ενώ της, της πολιτικής συνοχής πώς αντιμετωπίζουν τους διάφορους εξωτερικούς και ε, εσωτερικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, έχουμε πρόσβαση στις υποδομές αλλά, ε, από το Ταμείο Συνοχής, αλλά δεν αρκεί. Το ΕΤΠΑ προβλέπει και πρόσβαση στις υποδομές, αλλά και θέματα πληροφορικής και ε, κεφαλαίου. Αν καλύπτει και εξωτερικούς παράγοντες αλλά και εσωτερικούς όπως μεταβίβαση τεχνολογίας, εξωτερική θέση, ανθρώπινο κεφάλαιο και έχουμε πολύ ευρύτερο φάσμα. Το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας δεν προβλέπουν άμεση πρόσβαση, δικτύωση, ενημέρωση και τεχνολογίες πληροφορικής. Και αναφέρονται και στο ρυθμιστικό πλαίσιο διασυνοριακά. Ενώ το κοινωνικό ταμείο ε, αναφέρεται κυρίως σε διαχείριση δεξιοτήτων και στήριξη της αγοράς. Υπάρχει ένα μέσο, το Chessman, που προβλέπει πρόσβαση σε, σε κεφάλαιο και πληροφορίες και το Jeremy που επίσης απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιλαμβάνεται στα επιχειρησιακά προγράμματα και προβλέπει πρόσβαση στο κεφάλαιο, όχι στην υποδομή, λάθος, και στην πληροφορία. Τώρα, τι κάνει η πολιτική συνοχής και, το Ταμείο Συνοχής. Τι κονδύλια δαπανώνται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα επανέρχομαι σε κάτι πιο τεχνικό που είπα και πριν για τους κώδικες παρέμβασης. Αν προσθέσουμε ε, τους διάφορους κώδικες, φτάνουμε σε ένα μέσο όρο 68 δισεκατομμυρίων ευρώ που δίνονται για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή 20%, ένα πέμπτο των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής. Αυτά τα ποσά βέβαια διαφέρουν ανάλογα με το αν μιλούμε για τις 15 πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί έχουμε ένα τέταρτο του ποσού που αφιερώνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ στις νέες χώρες έχουμε ένα μέσο όρο 15% που δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Φιλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και κάτω χώρες, έχουν, δίνουν μεγάλη έμφαση σχεδόν το μισό ή και πάνω από το μισό δεκατό όλων των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι καθόλου αμεληταίο αυτό το ποσό. Μιλούμε για αρκετά δαψιλά κονδύλια. Τώρα, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε συγκρίση με την προηγούμενη περίοδο, γιατί αυτοί οι κώδικες παρέμβασης είναι κάτι καινοτόμο της νέας περίοδου και η εξπόστα αξιολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έδειξε ότι στην προηγούμενη περίοδο στι περιοχέ του στόχου 2, περιφέρειε του στόχου 2, τα μισά κονδύλια πήγαιναν στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και στι περιφέρειε του στόχου 1, 26%, δηλαδή ένα τέταρτο περίπου αφιερώνονταν στι μικρομεσαίες. Τι διδαχθήκαμε από το πώς καταφέρουν τα διαρθρωτικά ταμεία να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς επηρεάζουν τους δείκτες των επιδόσεών τους. Η προηγούμενη περίοδος μας έδειξε ότι δίνεται έμφαση στους δείκτες και δίνονται πολλές, ε, έμφαση δίνεται και συγκέντρωση πληροφοριών. Τι γίνεται με τις στρατηγικές εκθέσεις. Οι στρατηγικές εκθέσεις είναι εξαιρετικές και προσφέρουν διαφωτιστικές πληροφορίες ό,τι αφορά την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής συνοχής από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αυστριακή έκθεση, για παράδειγμα, δίνει πληροφορίες για output και τελικά αποτελέσματα και μιλάει και για τις δεσμεύσεις αναλήψεις υποχρεώσεων, αλλά λέει ότι οι δαπάνε και η αναλήψη υποχρεώσεων υστερούν σε σχέση με τους αρχικούς στόχους. Αυτό βέβαια είναι ένα γενικό φαινόμενο σε όλα τα κράτη-μέλη η έκθεση στρατηγικής και η Μαλτέζικη αναφέρονται άμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε άλλες χώρες οι στρατηγικές εκθέσεις δίνουν ελάχιστες πληροφορίες για το πώς οι επιχειρήσεις, όχι μόνο οι μικρομεσαίες, λαμβάνουν τέτοια κονδύλια. Το τσεχι... Η τσεχική έκθεση, για παράδειγμα, η τσεχική έκθεση στρατηγικής, δίνει αρκετές πληροφορίες για τη σχέση του προγράμματος με τις επιδόσεις την αποδοτικότητα, αλλά δεν μιλάει καθόλου για τις απο... επιδόσεις των επιχειρήσεων. Οπότε οι εκθέσεις στρατηγικής είναι τερόκλητες από αυτή την άποψη της παροχής τέτοιων στοιχείων. Οπότε δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συγκρίσιμα στοιχεία α, από τις εκθέσεις αυτές. Δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε δηλαδή με ποιο τρόπο η πολιτική συνοχή συνέβαλε στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το δίκτυο αξιολόγηση της Γενικής Διεύθυνσης ΡΕΓΚΙΟ προσπάθησε να εξαγάγει περισσότερες πληροφορίες από ε, τις ετήσιες έκθεσεις, ε, από τις εκθέσεις εφαρμογής και να συγκεντρώσει και άλλες πληροφορίες. Αναλύσαμε αυτή την έκθεση και στον πίνακα 15 της ε, μελέτης μας βλέπετε ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Εκεί έχουμε στοιχεία για επενδύσεις σε αποσχολήσεις, σε σχέδια ITT, σχέδια συνεργασίας και μερικά άλλα. Πολύ γενικοί δείκτες και ελάχιστα ένα τέταρτο των κρατών μελών δίνει τις πληροφορίες. Δηλαδή τρία τέταρτα των κρατών μελών δεν δίνουν καθόλου συγκρίσιμες πληροφορίες. Having said τούτων λεχθέντων. Αναλύσαμε 8 επιχειρησιακά προγράμματα, μπήκαμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αλλά και πάλι μόνο με βάση τις ε, πληροφορίες που δημοσιεύονται, τις αιτήσει δηλαδή, θέσεις εφαρμογής. Δεν πήγαμε στους διαχειριστές των προγραμμάτων. Επιλέξαμε λοιπόν 8 περιπτώσεις και δι' υποτίθεται πως είναι τα μεγαλύτερα προγράμματα που στοχεύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τον στόχο ανταγωνιστικότητας ε, κοιτάξαμε το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας, το πολωνικό πρόγραμμα και το ε, πορτογαλικό πρόγραμμα. Είχαμε τέσσερα προγράμματα περιφερειακής ανταγωνιστικότητας ε, και ανάπτυξης Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, ε, Ουγγαρίας, ε, Κεντρική Αγγλία και άλλη μια περιοχή, καθώ και ένα πρόγραμμα εδάφική ε, συνεργασία. Υπήρχε λοιπόν μεγάλη ποικιλία στο, στα κονδύλια που πηγαίνουν στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Το πολωνικό ήταν το μεγαλύτερο με 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ένα πολύ μικρό πρόγραμμα, ποσό βεβαίω για το πρόγραμμα τη Βαλτική. Τι μέτρα στηρίζουν αυτά τα προγράμματα, περί τίνος πρόκειται είναι πολύ διαφορετικά, πολύ Καλύπτουν από κουπόνια καινοτομία μέχρι επενδυτικά ταμεία, μέχρι ένα ταμείο για τον κινηματογράφο στην Πολωνία και τα οπτικοακουστικά μέσα. Είναι λοιπόν ευρύτατα. Και στοχεύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαφόρων τύπων όσον αφορά τα μέσα το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι πολύ, τα επιχειρησιακά προγράμματα είναι πολύ λεπτομερή και δίνουν αρκετές πληροφορίες για το τι μέσα είχαν. Ποιο ήταν ο στόχος μας το να μπούμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε αυτές τις ε, περιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να απαντήσουμε στο ερώτημα ε, του εάν αντιλαμβανόμαστε τις διαφορετικές διαστάσεις ε, της επίδοσης που σχετίζονται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εάν μπορούμε να αναλύσουμε το πώς οι διαχειριστικές αρχές αντιμετωπίζουν τα διαφορετικά προβλήματα. Και τι μαθαίνουμε από αυτό. Τι μάθαμε από αυτό. So, first of all, there... Πρώτα απ' όλα λοιπόν Υπάρχουν ε, διαφορετικές οικογένειες επιχειρησιακών προγραμμάτων. Να μπορούμε λοιπόν κάπως να γενικεύσουμε. Υπάρχουν εθνικά τέτοια προγράμματα που στοχεύουν ε, τις εθνικές ε, επιχειρήσεις και καλύπτουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό χρηματοδότησης. Είναι αν θέλετε μια ομπρέλα. Συχνά υπάρχει μια συμπληρωματικότητα καθώς και τα περιφερειακά προγράμματα στοχεύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άλλες φορές γίνεται μια διάκριση, αλλά τα εθνικά προγράμματα είναι αρκετά ε, εκτεταμένα και υπάρχουν κάποιες άλλες επικαλύψεις με τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Όμως, εάν δείτε τα περιφερειακά, προγράμματα ανταγωνιστικότητα, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ένα κλάσμα μόνο του συνόλου. Ένας, δύο άξονες προτεραιότητας. Μιλάμε για προσαρμοσμικότητα και μικρομεσαίε επιχειρήσει Αυτά είναι μικρό μέρος του προγράμματος. Και αυτό παρά το ότι έχουμε επιλέξει αυτά τα προγράμματα τα οποία έχουν τις μεγαλύτερες κατανομές για μικρομεσαίε επιχειρήσει. Τι βλέπουμε λοιπόν και θα ήθελα να προσπαθήσω να το περιγράψω. έχουμε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα Έχουμε έναν κατάλογο δαπανών ανακώδικα οπότε κατά κανόνα μπορεί να πει κανείς ε, ποιο ποσοστό των κονδυλίων πηγαίνει σε κάθε διαφορετική μορφή στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόβλημα είναι πως ε, παρά το ότι υπάρχει το σύστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδέσουμε αυτές τις δαπάνες με προτεραιότητες και μέτρα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε στα αλήθεια πώς η ποια κατανομή πηγαίνει σε κάθε προτεραιότητα και αυτό είναι μετά το πρόβλημα με τις αιτήσει εκθέσεις εφαρμογής. Γιατί οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής αναφέρουν σε βασικούς δείκτες και δείκτες στόχους, δεν αναφέρουν τις απάνες. Αυτή είναι μια γενίκευση, βεβαίως δεν ισχύει γιατί κάποιες εκθέσεις το κάνουν αυτό, κάποιες άλλες όχι. Οπότε το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορούμε να μετρήσουμε τις αιτήσιες δαπάνες ε, που σχετίζονται ειδικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό το οποίο είναι κάπως ανησυχητικό είναι πως τις αιτήσει αυτές τις εκθέσεις εφαρμογής υπάρχει αρκετά μεγάλος αριθμός δίκτων αριθμός ε, έργων ε, άμεσης στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αριθμός νέων επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν, αριθμός έργων ε, πληροφορικής. Οπότε, μετράμε τον αριθμό των έργων για να δούμε πώς στοχεύονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε λοιπόν αρκετές πληροφορίες όπου θα έλεγα πως είναι πληροφορίες που δεν μπορούν να μας πούν κάτι ουσιαστικό για το τι κάνουν τα ε, προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε δείκτες που είναι δύσκολο να κρίνουμε. Είναι πολλά, 300 έργα στην Πολωνία για ε, τηλεπικοινωνίες. Είναι λίγα, είναι πολλές πληροφορίες που μας δίνουν όμως λίγες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Αλλά πρέπει να πούμε που οι αιτήσεις εκθέσεις αυτές ε, δεν έχουν στόχο να απαντήσουν το ερώτημα που εμείς θέτουμε. Το είπα ήδη αυτό. Not a single of these common baseline indicators taking into account the SME situation. Πρέπει λοιπόν ε, να υπάρχει κάποια, ένα βασικό σημείο αναφοράς, να δούμε τι μπορούμε να πούμε σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βέβαια να ξέρουμε να κρίνουμε, να, να έχουμε ένα δίκτυο για να κρίνουμε αν κάτι είναι πολύ λίγο. Τι συμπεράσματα λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε. Έχω βγάλει έτσι συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν διαφορετική φύση. Ο ορισμός αυτός έχει μείνει λίγο πίσω που ισχύει. Όπως είπα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαφέρουν αρκετά. Οπότε για να έχουμε μια πιο στοχευμένη προσέγγιση Χρειάζεται μια πιο συνεκτική ανάλυση σε βάθος της μικρομεσαίας επιχείρησης, ε, στις διαφορές φάσεις της ζωής της, που να συμπληρώνει τον ε, τωρινό ορισμό. Το δεύτερο συμπέρασμα που βγάλαμε είναι πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδέουμε πολιτικές και μέσα με τους δείκτες αυτούς ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχοντας εξετάσει πολλά επιχειρησιακά προγράμματα και τη βιβλιογραφία είδαμε πως ε, οι χρηματοδοτικές αρχές έχουν μια γενικευμένη προσέγγιση για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπάρχει έλλειψη στρατηγικής και μια καθαρής λογικής σε εάν πάμε σε διάφορους κλάδους που θέλουμε να στηρίξουμε, σε φάσεις της ανάπτυξης, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, θα έχουμε... Θα έχουμε κάποια, βασικούς, κάποια βασικά συστατικά της πολιτικής αυτής. Οπότε, η πολιτική συνοχής, καθώς μάλιστα μιλάμε για αρκετά λεφτά τα οποία πηγαίνουν στους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να έχει μια συστηματική προσέγγιση ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται κάθε μικρομεσαία επιχείρηση και ειδικά και αυτό νομίζω πως είναι ένα από τα προβλήματα που προκύπτει από το ότι τα ταμεία συνοχής στοχεύουν συγκεκριμένες πολιτικές. Πρέπει να αντιληφθούν καλύτερα μια πολιτική μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να έχουν κάποιους στόχους. Το να γενικεύουμε δηλαδή τη μικρομεσαία επιχείρηση είναι ένα λάθος το να πηγαίνουμε σε διαφορετικές ομάδες στόχου. νομίζω πως είναι μια στρατηγική για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Ένα άλλο, μια άλλη σύσταση είναι οι στρατηγικές στήριξης να στοχεύσουν περισσότερο προς ε, τις δεξιότητες, στην καινοτομία και ανάπτυξη με έμφαση στα δύο τελευταία. Όπως είπα πριν, οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θέλουν να αναπτυχθούν και πολλές από αυτές δεν καινοτομούν και είναι επιτυχείς. Οπότε αν η πολιτική συνοχή έχει μια τόσο ευρεία προσέγγιση μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πρέπει να εστιάζει τόσο πολύ στην ε, καινοτομία και την ε, πληροφορική γιατί έτσι απομακρύνουμε πολλές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί η πολιτική αυτή είναι πολύ περίπλοκη. Επίσης κάτι προκαλεί εντύπωση. Τα μέσα της πολιτικής αυτής, ειδικά στα παλιά κράτη-μέλη, δεν συνδέονται πάντα με τα πιο σημαντικά τα κέντρα χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δεν σχετίζονται άμεσα με το τι χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και τα εθνικά μέσα. Υπάρχουν και επίσης τα ευρωπαϊκά μέσα τα οποία συνδέονται χαλαρά θα έλεγα με την πολιτική συνοχή. Και βεβαίω υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την πολιτική συνοχή και την προσβασιμότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ρητά αποφεύγουν το να ζητήσουν χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχή, από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ, σε τέτοια προγράμματα δηλαδή, πρώτα απ' όλα γιατί φαίνεται πως υπάρχει μία στάθεια στους κανόνες οι οποίοι αλλάζουν και δεν υπάρχει προχρηματοδότηση, ειδικά αν σκεφτούμε τις μικρές επιχειρήσεις, δεν μπορούν να προχρηματοδοτήσουν μόνες τους ε, για πολύ καιρό Οπότε υπάρχει αυτό το αίτημα να σκεφτούμε τις διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες θα είναι απλούστερες, να λάβουμε υπόψη πως οι μικροεπιχειρήσεις χρειάζονται δεξιότητες για να κάνουν την αίτηση για χρηματοδότηση, οπότε χρειάζεται κάποια αναλογικότητα στο τι πληροφορίες τους ζητάμε. Και βεβαίως μιλάμε για απλά πανάλ πράγματα. Τα έχουμε δει, είναι ε, δεξιότητες οι οποίες διαφέρουν σε κάθε αίτηση βεβαίω και κάθε αίτηση ζητάει διαφορετικές πληροφορίες. Αυτό το οποίο δεν είπα στην παρουσίασή μου, γιατί νομίζω πως δεν πρέπει να μακρηγορήσω κιόλα. The instruments that have been, let's say, put in place recently, they seem to have a fairly slow start. So I think είναι πως ξεκινάνε σιγά σιγά οι επιχειρήσεις. Νομίζω πως είχαν γύρω στις 30 ε, τέτοιες περιπτώσεις που είχαν δηλωθεί μέχρι το τέλος 2009. Είναι πολύ δύσκολο να λάβουμε τέτοιες πληροφορίες και αυτό φαίνεται να είναι ένα από τα προβλήματα των ε, ταμείων αυτών, καθώς ε, δεν υπάρχει, δεν κολλάνε πάρα πολύ με στρατηγική των διαρθρωτικών ταμείων. Και αυτό το οποίο μας ζητάνε για τις επόμενες ε, προγραμματικές περιόδους είναι να μην πάνε τα πάντα σε κυλιόμενα ταμεία, αλλά να υπάρχουν ε, και επιχορηγήσεις ειδικά για επιχειρήσεις οι οποίες ξεκινάνε. Και όταν ε, μιλάμε για τα διαρθρωτικά ταμεία και μηχανισμούς χρηματοοικονομικούς, το θέμα είναι ποιος διαχειρίζεται και πώς γίνεται η διασύνδεση. Η πολιτική συνοχή λοιπόν πρέπει να δίνει καλύτερα στοιχεία για το αποτέλεσμα και τον αντίκτυπο της στήριξη των επιχειρήσεων και θέλω να το τονίσω αυτό με βάση την ανάλυση της βιβλιογραφίας και τις 8 περιπτώσεις που είδαμε δεν είναι δυνατόν να δώσουμε στοιχεία για την επιτυχία ή μη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν ζητάμε η ε, παρακολούθηση ε, να δώσει αυτά τα στοιχεία γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ ποικιλόμορφες αλλά νομίζουμε πως θα ήταν χρήσιμο να ευθυγραμμίσουμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε όπως κωδικούς δαπανών με τις προτεραιότητες για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το υλικό το οποίο έχουμε αλλά να έχουμε πιο ποιοτικές και λοιπές ε, τεχνικές να δούμε παραδείγματο χάρη ε, αξιολόγηση τύπου και να δώσουμε περισσότερη σημασία στην αξιολόγηση του ζητήματος αυτού γιατί καλύπτει ένα 20% των δαπανών. Ναι, νομίζω τελείωσα με την παρουσίαση αυτή. Ήθελα να επίσης να σας στήσω την κυρία Χάμσα η οποία συνεισέφερε στη μελέτη αυτή και ευχαριστώ και την κυρία Ρούντολφ η οποία, με την οποία είχαμε έτσι, έντονες συζητήσεις για να καταλήξουμε σε αυτά τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θέλω να ρωτήσω τους συναδέρφους αν έχουν ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις. No. Would, would you like please to add something else or just finish now? Έχετε να μας πείτε κάτι άλλο ή έχετε ολοκληρώσει. In the case that we receive some questions. Σε περίπτωση που λάβουμε κάποιες ερωτήσεις θα σας τις αποστείλουμε με το ταχυδρομείο. Για μια φορά ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό είναι το πέρας της συνεδρίασης. Ευχαριστώ.